Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Allons-y. Nous allons ouvrir. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ε, θα αρχίσει η συνεδρία σας σιγά σιγά. Ε, αλλά προηγουμένως, αγαπητοί συνάδελφοι, Πριν αρχίσουμε έλεγα τις εργασίες τη Επιτροπής, θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω eh oui, ε, τον κύριο Κώστη που ε, κάθεται εδώ αριστερά μου είναι η τελευταία μέρα σήμερα Πρέπει να το χειροκροτήσετε ε, ταυτόχρονα όλοι τον Κωστή. Φεύγει από τη γραμματεία ο Κωστής. Θα πάει προς άλλους ορίζοντες, σε άλλα νερά που ονομάζονται γραμματεία Ήτρε. Δεν ξέρω αν είναι πιο συμπαθής από εμά, δεν νομίζω. Πέντε χρόνια ήταν στη γραμματεία μας για πολύ σημαντικά θέματα. Είτε ήταν το συνδρομικό πακέτο, τη λευκή βίβλο ε, για τις μεταφορές ή ε, την βαγγίσεως των μεταφορών από το διοξίδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ Κωστή. Ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ελπίζω και στην Ήτρα να τα πάτε τόσο καλά όσο και στην Επιτροπή Μεταφορών. Πάντως η πόρτα και της Γραμματείας και της Επιτροπής μας θα παραμένει πάντα ανοιχτή για σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με θέματα πιο πεζά. Ε, θα ε, ελέγξουμε τα μηχανήματα. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τις κάρτες για να δούμε αν είναι παρόντες όσοι βουλευτές πρέπει από κάθε ομάδα. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est fermé. non. C'est très Πολύ ωραία. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, ειλικρινά, αλλά νομίζω ότι ξέχασα στο Στρασβούργο την κάρτα ψηφοφορία μου. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διακτηνιστώ. Θα προσπαθήσω να τη βρω κάποια στιγμή. Τώρα πώ θα το λύσουμε αυτό. Καταρχά, σα ζητώ συγγνώμη. Alors, comment... Λοιπόν, Πώς θα το χειριστούμε αυτό. Πολύ απλά. Θα σηκώνετε το χέρι σας. Υπέρ κατά αποχή. Και θα καταμετρηθεί κάθε φορά η ψήφος. Ωραία. Συμφωνείτε. Πάμε λοιπόν. Έχουμε πολλές ε, ψηφοφορίες σήμερα. Κύριε Τέιλορ. Καλημέρα σας. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Στέλλερ. Δεν λειτουργεί η κάρτα σας. Τι λέτε κύριε Ρίκια, για Brexit πρωινιάτικα 9 η ώρα το πρωί. Αφήστε το. ωραία. Τώρα είναι εντάξει. Προχωρούμε. Πρώτη ψηφοφορία έκθεση του κυρίου Τέλιτσκα. Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Αρχίζουμε. Συμβαστική πρώτη Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία υπερθών 1. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Απόχες Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 36 υπέρ. Qui est Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 38 υπέρ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 αποχές η τροπολογία 6 δεν εγκρίνεται η τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8. Συμβαστική 9 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, παρακαλώ. J'ouvre le vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Το ΕΛΚ έχει δύο παρακαλώ υπεράριθμους. Καλά, ένα πάει και έρχεται, αλλά δύο το παρακάνετε. Κλείνει η ψηφοφορία. Alors, plus 19. 19 υπέρ, 24 κατά, η τροπολογία απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Όχι, ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, την 84 ψηφίζουμε τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, έτσι δεν είναι. Θέλετε πολύ Ωραία. Πολιθεύουμε την τροπολογία 4. 84 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 29-15. Συνεχίζουμε. Συμβαστική 10 ψήφι πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 99 ΕΠΕ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 ΕΠΕ Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 ΕΠΕ Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 ΕΠΕ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 19 συμβαστική υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα θα θέσω προς ψήφιση το σύνολο ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και τελειώνει. 43 υπέρ, ένας ε, κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Τέλιτσκα, ε, κρίθηκε η έκθεσή σας. Καλά, δεν πειράζει, χειροκτοτήστε το. Allez, nous continuons. Encore avec vous, monsieur. Συνεχίζουμε. Πάλι δική σας έκθεση, κύριε Τέλισκα, σχετικά με τα πρότυπα. εφαρμογή κανονισμού. Amendement 2. Πάμε λοιπόν, τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 και 4 ε, ταυτίζονται υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Απόρριψετε. Η συμβαστική έξι Τσεκ φωνές από κάτω. Ωραία. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην 23. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Πάλι περσεύει ένας από το ΕΛΚ. Πολύ δραστήριο σας βρίσκω.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 58 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τσεκ, ωραία. Αρχίζει η ηλεκτρονική παλήθευση. Τώρα αρχίζει δηλαδή. Τα γνωστά, από το ΕΛΚ πάντα ένας υπεράριθμος. Τώρα είμαστε εντάξει. 23 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν το πρώτο τμήμα, όπως είπα. Δεύτερο τμήμα, ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται το δεύτερο. Συμβαστική 12. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία αριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Le vote est clos. Πέρας. 43 υπέρ, ένας αντίθετος και μηδέν αποχές. Εγκρίνεται η έκθεσή σας. Και πάλι κύριε Τέλιτσκα, σε Allez, nous continuons. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την έκθεση για την εγγραφή των επιβατών στα επιβατικά πλοία που εκτελούν δρομολόγια, έκθεση Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, με συγχωρείτε. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πολλές πολλές ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 48 υπέρ κατά Αποχές. Η 48 απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 49 εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε απευθείας στην 51. Είναι ταυτόσιμες. 13 πρώτα και, 15, και 52 μαζί που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Και τώρα Περνάμε απευθείας στη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν αγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 59 εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, η 60 απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, η 2 εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, η 55 απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές η 66 απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές 67 εγκρίνεται μου φαίνεται θέλετε να κάνουμε επαλήθευση έλεγχος λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. 68 υπέρ, κατά, αποχές. 68 εγκρίνεται. Καταπίπτουν γιατί εγκρίθηκε 68. 71 υπέρ, κατά, αποχές. Η 71 απορρίπτεται. Είμαστε στην τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές η 73 απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές η 19 εγκρίνεται 75 υπέρ Κατά. Αποχές. Η 75 απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 78 απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 79 εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές. Η 21 εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές. Η 22 εγκρίνεται. Περνάμε σε ταυτόσιμες τροπολογίες. Η 84 και η 83. Υπέρ κατά αποχές αυτές οι δύο τροπολογίες απορρίπτονται 85 και 86 τώρα Α, θέλετε επαλήθευση 83-84, ωραία Άρχεται η ψηφοφορία Η ψηφοφορία έληξε Συν 20, 25 Μηδέν αποχές, άρα απορρίπτονται Συνεχίζουμε. 85 και 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτές οι δύο τροπολογίες απορρίπτονται. Όχι, απορρίπτονται. Απορρίπτονται καλά καλά. Θέλετε παλήθευση. Άντε. Εντάξει λοιπόν. 85 και 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Ναι, το ίδιο. Συν 20 μείον 25. Απορρίπτονται ξεκάθαρα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 23. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 και 26 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 25 υπέρ κατά αποχές ή 25 εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές η συμβαστική 4 εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 4 και 29 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πάμε απευθείας στην 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 33 εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 34 εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 35 απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές η συμβαστική 5 εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές η 39 απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές η 40 απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές η τροπολογία 6 7 υπέρ. Κατά αποχές η 7 εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές η 8 εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται. Πέρας. 44 υπέρ, καμία ψήφο κατά και καμία εποχή. Μπράβο σα κύριε Μπαραντίκα. Α, μία ψήφο κατά. Ναι, ξέχασα, ξέχασα δεν είχατε την κάρτα σα. Μπράβο σα κύριε Μπαραντίκα Μπιλμπάου. Και τώρα θα ψηφίσουμε και για την εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Υποτακτική εντολή. Πέρας. Συν 43. Μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Έχετε διαπραγματευτική εντολή για αυτή την έκθεση. Μπράβο σας. Πάμε, συνεχίζουμε με το σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων μοχηματαγωγά ρορό και ταχύπλε επιβατηγά σκάφη, έκθεση του κυρίου Ρικέ. Πάμε. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε απευθείας στην 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 22 εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. Κυρία Φώστερ, Ψηφίζουμε συγκέντρωση. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές η 8 εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές η τροπολογία η τροπολογία 9 εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά Αποχές. 25 εγκρίνεται. 10 υπέρ. Θέλετε να κάνουμε παλήθευση. 25. Εντάξει λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 ε, υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 10 υπέρ, κατά, αποχές, η 10 εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, η 11 εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, η 26 εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, η 27 εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές η 29 εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές η 30 εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές η 31 εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές η 1 εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές η 13 εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές η 14 εγκρίνεται. 15 υπέρ. 15 υπέρ. Κατά αποχές η 15 εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές η 17 εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Η 18 εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζεται όλη η έκθεση. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 45 ψήφοι υπέρ, καμία ε, ψήφος κατά, καμία εποχή. Α, υπάρχει μία ψήφος κατά και καμία εποχή. Κύριε Ρικέ, μπράβο σας. Και τώρα δεύτερο σκέλος, να ψηφίσουμε και για τη δημοκρατική εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 44 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμιά αποχή, η διαπραγματευτική εντολή εγκρίνεται, κύριε Ρικέ. Μπράβο σας. Και τώρα συνεχίζουμε. Με την έκθεση της κυρίας Αγιούτο. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατικά πλοία. Πάμε να ξεκινήσουμε. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. 39 και 40 ταυτόσιμες. Υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται άρχεται η ψηφοφορία πέρας συν 25 μείον 20 άρα εγκρίνεται να με συγχωρείτε καλά καλά και ζητήσατε επαλήθευση 41. Υπέρ. Κατά. Αποθέσω. Δεν εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Η συμβαστική δεν εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 43 απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Θέλετε έλεγχο. Κανένα πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφοφορία για την τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συν 13 με 28. Απορρίπτεται. Δεν είπα απορρίπτεται καλά καλά, είπα απορρίπτεται απλώς. Κύριε Αρτούκ, ναι μήπως θα μπορούσαμε να περιμένουμε δύο δευτερόλεπτα. Διότι η διερμηνία είναι λίγο πιο αργή από τη δική σας η εκφώνηση των αριθμών των τροπολογιών. Καλά, θα περιμένουμε λίγο περισσότερο. Θα είμαστε λίγο πιο αργοί. Πάμε. 43 απορρίπτεται. 4. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές η 4 εγκρίνεται συμβεβαστική 3 ποιος είναι υπέρ ποιος είναι κατά αποχές η 3 εγκρίνεται 49 υπέρ κατά Αποχές. Η 49 εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 13 δεν είμαι βέβαιο ότι εγκρίνεται. Σηκώστε καλά το χέρι. Α, έρχεται η ψηφοφορία. Για τη 13 μιλάμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, εγκρίνεται. Και μάλιστα ξεκάθαρα. Δεν σηκώνεται αρκετά τα χέρια. Λοιπόν, 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 14 δεν νομίζω να εγκρίνεται. Αλλά θα επαληθεύσω. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την τροπολογία 14. Πέρας. Η 14 δεν εγκρίνεται. 25 ψήφι κατά, 20 υπέρ. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. 56 ε, απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. 57 ε, απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. 58 ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. 15 εγκρίνεται. 59 υπέρ. Με συγχωρείτε, 59 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 59 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 59 θέλετε παλήθευση. Να ανοίξω τη ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 59. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, Συν 25 μείον 20. 25 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το δεύτερο τμήμα δεν απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, η τοπολογία 2 εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, η τροπολογία 3 εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, 26 νομίζω δεν εγκρίνεται. Αλλά θα ελέγξουμε. 26 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, εγκρίθηκε. Συν 32, μείον 13. Η 26 εγκρίνεται καλά καλά. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές η συμβαστική αναγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απευθεία συμβαστική 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές ή 32 εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Παρακαλώ. Πέρας. 45 ψήφι υπέρ. 46, 46 ψήφι υπέρ, καμία αποχή. Και καμία ψήφος κατά. Κυρία Γιούτο, μπράβο σας. Νομίζω ότι αποτελεί ρεκόρ για την ε, Επιτροπή μας. Εγκρίθηκε η έκθεσή σας. Και τώρα φυσικά θα ψηφίσουμε την διαπραγματευτική εντολή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 45 υπέρ, μία ψήφος κατά. Έχετε και τη διαπραγματευτική εντολή για να συνεχίσετε τις συζητήσεις θέμα του θέματος. Κυρία Γιούτο, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε. Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Συνεργατική Οικονομία είναι το επόμενο θέμα. Σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΝΚΟΕ, συντάκτρια κυρία Κίλονεν. Κοιτάξτε, έσυ λίγο ηρεμία, σας ακούμε μέχρι εδώ τους συμβούλους. Λοιπόν, συμβιβαστική ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, προτιμώ να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 20. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή και άλλη μία κατά. Εγκρίνεται τροπολογία. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 4. Τροπολογία 50. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ελέγχουμε. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 7 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 68. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 68. Τροπολογία 69. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, δεν γίνεται δεκτή, αλλά δεν συμφωνείτε να το ελέγξουμε. Στην 72 είμαστε. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ. 8 κατά. Με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται. Λοιπόν, περνάμε συμβαστική 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 75. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 και 96 ταυτόσμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 91 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε, δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 91. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψηφί υπέρ, 20 κατά. 20, μία κατά. Άρα εγκρίνεται. Η 91 και περνάμε στην 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 129. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές αποχές να ελέγξουμε καλύτερα θα έλεγα. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 22 κατά. Είχα δίκιο, εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία έρχεται Ψήσατε όλοι πέρα στις φοφορίες. 39 υπέρ, 7 κατά, δεν υπάρχει αποχή. Η κυρία Κίλων την εκθεσή σα. Σα ευχαριστούμε. Allez, nous Συνεχίζουμε. Προαγωγή τη σύνδεση των διαδίκτυων στι τοπικέ κοινότητε είναι το επόμενο θέμα. Σχέδιο γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Ήτρε με συντάκτρια την κυρία Ταπαρδέλ. Φύγαμε. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 55. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ. 23 κατά. Καλά έκανα και έλεγξα. Διότι απορρίφθηκε η τροπολογία. Συμβεβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Τροπολογία 65. Πέραση ψηφοφορίας. Κύριε Βαντεκάμπ, σε φες. Απορρίφθηκε η τροπολογία. 66 ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβα... μάλλον συγγνώμη τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 6. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογή 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογή 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ξαναρχίζουμε. Τροπολογή 27. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 27. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβεβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 12 η συμβιβαστική. Θέλετε να το ελέγξουμε όμως. Να ελέγξουμε τη συμβιβαστική 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Συνεχίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελειώσαμε. τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 44 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται σα και τα παρδέλης χαρητήρια. Συνεχίζουμε. Έκθεση για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα, για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabit και του 5G. Σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Ήτρε από τον κύριο Ζλοτόφσκι. Τώρα το είπα καλά. Δεν έχετε παράπονο. Το είπα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική α, α, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε κατευθείαν στην τροπολογία 12, ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτη 14. Συμβιβαστική Β. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ. 33. Την έχετε. Λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική C υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. που πηγαίνουμε, στην 39 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική D, δέλτα, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά, αποχές η 53 εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογική 76. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Προπολογή 78 ψήφι ΠΕΡ. κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα η ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία άρχεται παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας 40 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Ποιο είναι, Ποιο ήταν? Α, ο κύριο Λοτόσκι ήταν. Μπράβο σας κύριε Λοτόσκι. Εγκρίνεται η έκθεση. Με πολύ ωραία πλειοψηφία. Κουράγιο. Μία μας έμεινε και είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Εδώ έχουμε τώρα την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τι απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τι υπηρεσίε. Και γνωμοδότηση για την Επιτροπή ΙΜΚΟ με συντάκτο κύριο Κιφ Τέιλορ. Φύγαμε. Τον τίτλο 1 πρώτα απ' όλα. Έχουμε τις τροπολίες από 31 έως 2.36 από κοινού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 129. Τι θέλετε, να ελέγξουμε τη συμβαστική 9, να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 22 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. παρόλα αυτά εγκρίνεται όπως είχα πει. Η συμβιβαστική να συνεχίζουμε με την τροπολογία 129. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 129 εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές ή 10 εγκρίνεται. 130. Καταπίπτει. Όλα αυτά καταπίπτουν. Συνεχίζουμε. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 132 απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 141 απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 12 απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. 144 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 146. Θέλετε έλεγχο. Καλώς. Αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην 145. Τέλος. 18 υπέρ 26 κατά. Έχετε δίκιο. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 146 τοπολογία. ψηφίπε. Κύριε Βέρνερ και κύριε Βάντενκαμπ. Για να συνταχθείτε λίγο παρακαλώ. Είναι τελευταία ψηφοφορία, λίγη υπομονή κάντε. 146 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 152. Καταπίπτει διότι εγκρίθηκε η προηγούμενη. 147 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 149 εφέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 150 εφέ. κατά άποχες απορρίπτεται 151 μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ με μεγάλη μου χαρά Άμα το ζητάτε τόσο ευγενικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. 150. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. 17 υπέρ 18 μάλλον 28 κατά απορρίπτεται η τροπολογία αυτή. Πρόεδρε, επειδή απερίφθη, θέλω να θέσω ένα διδικαστικό, αν δεν σας πειράζει, ως εξή. Η Επιτροπή καταψήφισε την τροπολογία μας 150 Ε, υπάρχει ε, συνεπής αναφορά στο τι εστί καταναλωτής και εσείς το καταψηφίσετε. Υπάρχει ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το τι εστί καταναλωτής. Είναι δύο τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο είναι φυσικό πρόσωπο και β, όταν συνάπτει μία σύμβαση, προχωρεί σε μια δραστηριότητα εκτός της εμπορικής ή επαγγελματικής του. Η δική μας λοιπόν ε, τροπολογία έχει το σωστό ορισμό. Κύριε Βουλευτά, αγαπητοί συνάδελφοι, τι διαδικαστικό είναι αυτό, καμία σχέση με τον κανονισμό δεν είμαστε εδώ για να συντάξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Δεν λαμβάνω υπόψη την παρατήρησή σας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε λέξεις την ώρα που ψηφίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η τροπολογία 150 λοιπόν απερίφθη. Η 151 ψηφίπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 επέ, κατά αποχές εγκρίνεται. Alors, nous n'avons... Alors, c'est la... Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αγγλική διερμηνία. Ε, τώρα είναι εντάξει. Παρακαλώ, ανοίξτε μικρόφωνα στην καμπίνα παριθμό 2. Non, non, ce n'est pas un coup du Brexit. Δεν φτάει το Brexit. Δεν επιτρέπω τέτοια σχόλια στην Επιτροπή μου. Λοιπόν, προχωρώ. το 13 Ouais. 10 Les techniciens. Λοιπόν, παρακαλούμε του τεχνικού. Υπάρχει θέμα και με τη φιλανδική διερμηνία. Αριθμό 10, λέει η κυρία Κίλονεν. Τώρα εντάξει. Ωραία. 151 εγκρίθηκε. 153 επίσης. Είμαστε στην 154 κύριε Βαντενκάμπ. Ψηφίπε. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Ψηφίπε. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 13. Υπέ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 164 ψήφι υπέ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 ψήφι υπέ κατά άποχες απορρίπτεται. 166. Θέλετε έλεγχο, παρακαλώ, για την 165 αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 165 εγκρίνεται. 28 υπέρ, 17 κατά. 18. Εγκρίνεται λοιπόν η 165. Το συγγνώμη, σωστά ζητήσατε παλήθευση. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Χρειάζεται και αυτό έλεγχο. Την 68 λέει η πρόεδρος, αλλά είναι 166. 166 διορθώνει. Πέρα. 28 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 175 ψήφι κατά Α, μάλιστα. Πού είναι η συμβαστική 15, γιατί στη στο δικό μου κατάλογο δεν το βλέπω και το θεώρησα ότι είναι τροπολογία απλή. Δεν είναι με έντονους χαρακτήρες, οπότε δεν την είδα. Άρα λοιπόν πάμε στη συμβαστική 15. Υπέ Κατά. Άποχες. Επαλήθευση παρακαλώ για τη συμβαστική 15 γιατί δεν ήταν σαφές. Πέρασε. 24 υπέρ 21 κατά εγκρίνεται η συμβαστική 15. Συνεχίζουμε. Η τροπολογία 175 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 ε, ε, με 182 υπέρ κατά άποχες Εγκρίνονται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Είναι 185. Τώρα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πέρας. Plus 12, moins 33. 12 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. Παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια σας. Τροπολογία 186 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά υπέρ ξανά παρακαλώ σηκώνετε χέρια α έτσι σας θέλω κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχο θέλετε παρακαλώ στην 187 23 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Ψηφί Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Πάμε πάλι λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία και τελειώνει τώρα. 31 υπέρ 14 κατά εγκρίνεται η συμβαστική. 189 μισό λεπτό καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η συμβαστική 16. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 193 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά άποχες απορρίπτεται 210 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται τσεκ ωραία το τσεκάρουμε 210 παρακαλώ αρχή ψηφοφορία λίγη τώρα 22 υπέρ, 24 κατά απορρίψετε. Συνεχίζουμε. 211 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 2.14 είπε, κατά άποχες εγκρίνεται 215 είπε, κατά άποχες απορρίπτεται 216 είπε, κατά άποχες εγκρίνεται 217 είπε. κατά άποχες εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ένας. 26 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Και είχατε δίκιο. Τροπολογία 222. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία, να επαληθέσουμε τη 222. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τη 222 εγκρίθηκε. 223. Ψήφι πέ Κατά. Αποχές. Αυτή απορρίπτεται 223 με μεγάλη διαφορά. 224 υπέ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225 υπέ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 233. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. στη συνέχεια. Όλο το παράρτημα 1 με όλες τις τροπολογίες αυτές που βλέπετε. 2.37, 2.40, 42, 46, 48 και 50. Υπέ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η συμβιβαστική μόνο 21. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε γυρίστε πολλές σελίδες τώρα. Και ε, βρισκόμαστε στην τροπολογία 258. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 260. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στη συνέχεια όλες τις τροπολογίες του παρτήματος 1 τμήμα 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3.33 και 3.62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3.63 ψηφί υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Η τοπολογία 364. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τοπολογία 30. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ξανά. Υπέρ της 30. Έτσι πράγμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 368 και 69 και 70. 3. Δεν είναι τη λογική σκέψη, είναι στο παράρτημα 1, τμήμα 10. Λοιπόν, 368, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η 368. 369 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε παρακαλώ. Είστε στην 369 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται 17 υπέρ 27 κατά. Η τροπολογία 370 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ακολουθούν τώρα οι υπόλοιπες τροπολογίες, η 33 είπε κατά άποχες εγκρίνεται. 34 είπε κατά άποχες απορρίπτεται. 35 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ φωνές. Αρχίζει η παλήθευση. 41. Πέρασε. 21 υπέρ 22 κατά. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ κύριε Βαντενικά που ζητήσατε παλήθευση. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται. Η 48. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, παρακαλώ. Άρχιτε ψηφοφορία στην 50. Je ferme le Πέρας. 21 υπέρ, 23 κατά. Είναι πολύ μικρή η διαφορά. Παρ' αυτό δεν εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52 ψήφι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 57 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 58 ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 6 ψηφί Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 59 Υπέ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 60 ψηφί Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 62 Υπέ. Κατά. Απόχες. Δεν εγκρίνεται 62. Τσεκ, φωνές, θέλετε έλεγχο, ωραία, μάλιστα. Ελέγχουμε τότε. Αρχίζει η πληροφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 18 κατά, είχατε δίκιο, εγκρίθηκε. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 65 Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι υπορρίπτεται αλλά προτιμώ να επαληθεύσω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ. 21 υπέρ, 23 ε, κατά. Γιατί είναι και εκεί μια ψήφος. Δεν εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική 3. Υπέρ. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μα δεν ψηφίσετε. χιτιέστε μεταξύ σας. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε έτσι, αλλά άντε, σε επαληθεύσουμε πάλι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Α, 21 υπέρ. 22, 23. Για μια ψήφο διαφορά. Δεν εγκρίνεται, δηλαδή απορρίπτεται. Οπότε θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες μία-μία. 68. Κατά. Θα κάνω επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 υπέρ 20 κατά. 69 ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία πάλι. Πέρας για την 69. 22 υπέρ. 22 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά. Συμβαστική 4 εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά προτιμώ να επαληθεύσω. Κάνουμε έλεγχο. Συμβαστική 5. Πέρας. 21-21. Α, 22 κατά. Ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες της συμβαστικής 5. Μία-μία. Γιατί δεν εγκρίθηκε η συμβαστική 5. Για να ξεκινήσουμε. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Θέλετε παλήθευση. Ωραία. Για την 7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι 84 εγκρίνεται, αλλά προτιμώ να επαληθεύσω. Άρχια την ψηφοφορία για την τροπολογία 84. Πέρας. 22 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές η 79 απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση. Να ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 79. Πέρας. «24 κατά, 20 υπέρ». Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Α, 80. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κατά τη δική μου την άποψη απορρίπτεται 80. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 82 απορρίπτεται. Συνεχίζουμε κανονικά. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 85 απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 87 εγκρίνεται. Πιστεύω. Θέλετε επαλήθευση να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 87. Πέρας της ψηφοφορίας. Συν 22. Μείον 22. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 89. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. 90 υπέρ. Α, καταπίπτει, να με συγχωρείτε. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 91 απορρίπτεται. 92 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 92. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 6 εγκρίνεται. Η 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. 98 εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 100 εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 102 απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 103 εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, ή 105 απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές, ή 106 εγκρίνεται. Εντάξει, τουλάχιστον παρακολουθείτε. Καλό αυτό. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 108 Απορρίπτει. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η 109 απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 110. Ψηφίζουμε το τελικό σχέδιο έκθεση όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται αυτή. Άρχεται. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ καμία αποχή μείον, όχι, 20 ε, εποχές καμία ψήφους κατά. Η έκθεση Τέιλορ εγκρίνεται. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Εντάξει, ωραία. Μία ψήφος κατά. Θα το γράψουμε στα πρακτικά. Μετά από αυτήν την εντατικότατη φάση ψηφοφοριών, θα διακόψουμε για 5 με 10 λεπτά την συνεδρίαση για να αφιχθούν οι προσκεκλημένοι μας. Α, βα, ήταν σαν.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

Mes chers collègues, nous allons reprendre notre... Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μα. Και έχουμε μεγάλη ακρόαση τώρα με θέμα γυναίκες και ο ρόλος τους στις μεταφορές για να επιληθεί το πρόβλημα ε, έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στις μεταφορές. Αποφασίσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε την παρούσα ακρόαση έτσι ώστε να ασχοληθούμε με το θέμα του φύλου ε, στις μεταφορές και να αναλύσουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό γυναικών που εργάζονται στις μεταφορές. Η ε, συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα ε, τα επόμενα χρόνια. Έχουμε εμπειρογνώμονες προσκαλέσει που καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας και θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε ε, με διάφορες πτυχές του θέματος, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, για την ισότητα των φύλων και πώς εφαρμόζει τις μεταφορές, ποια είναι η εμπειρία των κρατών μελών και συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στις μεταφορές καθώς επίσης και ε, από τη σκοπιά των ε, μεταφορικών επιχειρήσεων και πώς ε, προσλαμβάνουν και απασχολούν γυναίκες. Έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε για να ακούσουμε την αυτή εξοχότητα, την μόνιμη αντιπρόσωπο, αναπληρώτρια καλύτερα, της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία ε, πρέσβη ε, Αόσα Βέμπερ. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζιλ Μπεργκό. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Καθώς επίσης και εκπροσώπους του κλάδου. Την πολιτική γραμματέα ε, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταφορές, ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές, η κυρία Τίλινγκ, καλώς ορίσατε, καθώς επίσης και τη Γενική Γραμματέα της Ένωσης Ευρωπαϊκών που είναι η κυρία Χακστάινερ. Χακστάινερ. Μάλιστα. Καλώς ορίσατε. Alors, je voudrais que... Στην Επιτροπή μας. Κάθε μία από τις ομιλήτριές μας, γιατί ομιλήτριες έχουμε σήμερα, ε, έχετε ένα πεντάλεπτο και βέβαια στην πλειονότητα τους ε, οι κυρίες, έχουμε και τον κύριο Περζό, να, για να εξετάσουμε λοιπόν το θέμα του φύλου. Στις εργασίες μας και τα εισαγωγικά σχόλια θα κάνει ο εισηγητής μας, ο κύριος Νίλσον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Pour 5 minutes. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σου ειδικά σήμερα και θέλω να την αξιοποιήσω. Παρακαλώ να βάλετε ακουστικά για να μπορέσετε να με καταλάβετε. Είμαι μόνιμος εισηγητής ε, για αυτό το θέμα, αλλά έχω σειρά ετών εμπειρία στη Σουηδία, στην ε, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση για το θέμα του gender mainstreaming, δηλαδή την ε, ένταξη της έννοιας του φύλου στις διάφορες πολιτικές. Δεν καταλαβαίνουμε πάρα πολλές φορές τι σημαίνει αυτό. Για να το κατανοήσουμε δεν πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία. Ήδη ε, κατά τη δεκαετία του 90 στη Σουηδία αποφασίσαμε ότι το θέμα δεν είναι να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών γενικώ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρέπει να είναι η συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας που θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε να επέλθει ισότητα μεταξύ των φίλων. Πρόκειται για ίσα δικαιώματα προφανώς αλλά και για μια κοινωνία που θέλουμε να δημιουργήσουμε η οποία θα μετεξελίσσεται και θα επιθυμεί να μετεξελίσσεται. Διότι οι γυναίκες ε, θα πρέπει να αξιοποιούνται και αυτές στο έπακρο. Ε, δεν μπορούμε να αφήνουμε στην άκρη κάποιες δεξιότητες και ικανότητες γιατί δεν προχωράει έτσι η κοινωνία. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το gender mainstreaming. Εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών καταρτήσαμε στρατηγική πριν από λίγα χρόνια για το συγκεκριμένο θέμα και είχαμε πει ότι ε, θα πρέπει να ορίσουμε σαφείς προτεραιότητες. Αυτό ε, από τη μία έχει να κάνει με την κατάρτιση, με την, με την εκπαίδευση να έχουμε και σαφείς στατιστικές και συγκεκριμένες και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ε, αρμοδιότητα. Ε, θα πρέπει να έχουμε και περισσότερες γνώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των μεταφορών, γιατί αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. Ε, πρέπει να αποκομίσουμε μια καλύτερη εικόνα για την κατάσταση του κλάδου των μεταφορών. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη σημερινή μας ακρόαση. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνεργαζόμαστε με τους εργοδότες και σε μεγάλες και σε μικρές πόλεις. Έχω συνομιλήσει με έναν εκπρόσωπό τους που μας είπε εμείς θέλουμε καλούς οδηγούς. Δεν μας ενδιαφέρει είναι άνδρες ή γυναίκες. Και έχουμε καλούς οδηγούς στην εταιρεία μας. Αλλά πάντα είναι καλό να έχουμε ένα μείγμα. Είναι πάντα θετικό στην αγορά εργασίας, στον τόπο εργασίας να εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα. αν θέλουμε για λόγους οικονομικούς να προωθήσουμε την οικολογική οδήγηση, χρειάζονται και γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη επίγνωση ε, των συνεπειών ε, για το περιβάλλον και προσπαθούν να οδηγούν συνετά οικονομικά για να εξοικονομούν και καύσιμο. Ορίστε μια θετική επίπτωση στις μεταφορές από τη συμμετοχή των γυναικών. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλωσορίσω θερμά και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τι έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νίλσεν. Θέλω να σας πω ότι και η Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Απασχόλησης ε, συμμετείχαν στην Επιτροπή αυτή. Είναι συνδεδεμένη στην όλη διαδικασία. Δεν θέλω να δώσω, μάλλον δεν θέλω να μακρηγορήσω εγώ και να χάσουμε άλλο χρόνο. Έχετε ε, εσείς ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που είστε και στη μειονότητα ως φίλο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Έχετε 10 λεπτά για να μας διαφωτίσετε για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω που σκεφτήκατε να προσκαλέσετε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση αυτή για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Για να σας υπενθυμίσω αρχικά ποια είναι τα βασικά, δηλαδή ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένη στο πλαίσιο των συνθήκων, αλλά και από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται αυτή τη διάσταση του φύλου να την ενσωματώσει στις πολιτικές που αναπτύσσει. Φυσικά, πρόκειται για μια οριζόντια πολιτική Έχουμε τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών που καλύπτει την περίοδο 16-19 αρμοδιότητα της Επιτρόπου Γιούροβα και των υπηρεσιών της Δέλτα Just. Σήμερα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ε, ιδιαίτερη κατάσταση του τομέα των μεταφορών. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπενθυμίσω ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί για μας μεγάλη προτεραιότητα. Σε μεγάλο βαθμό, λόγω και της προσωπικής δέσμευσης ε, της ε, ε, Επιτρόπου μας, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και πρέπει να φέρουμε σε πέρα συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Έχουμε ήδη δρομολογήσει συγκεκριμένες δράσεις αληθεύει ότι στον τομέα των μεταφορών πολλή δουλειά πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πράγματα ακόμη που εκκρεμούν η κατάσταση γενικώ. Δεν είναι τόσο θετική σε σχέση με τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι γυναίκες είναι το 22 περίπου της 100 των απασχολημένων στον τομέα των μεταφορών ε, αυτή τη στιγμή σε σχέση με το 46% ε, στη γενική οικονομία και βέβαια η κατάσταση ε, ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς ε, και τη θέση. Δηλαδή σε τεχνικές επιχειρησιακές θέσεις ε, εκεί έχουμε τα χαμηλότερα σκορ ε, πολύ, μικρές, πολύ μικρά ποσοστά στις γυναίκες μηχανοδηγούς μόνο 3% άρα πάρα πολλά ακόμη πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό και η γενική απασχόληση πρέπει να σας πω ότι αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδιά για να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού που παρατηρείται ήδη στον τομέα των μεταφορών και το οποίο θα επιδεινωθεί στα επόμενα χρόνια. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ένα τρίτο των εργαζομένων σήμερα είναι πάνω, των, πάνω από 50, άρα θα βγουν σε σύνταξη σε λίγα χρόνια. Και από την άλλη είναι και οικονομικό πλεονέκτημα, γυναική απασχόληση, η οικονομική κλάδη, όπως είπαμε, που η ε, σχέση ανδρών και γυναικών είναι ισορροπημένη, είναι και οι τομείς όπου έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Έχουμε τώρα στις συγκεκριμένες δράσεις ε, που έχουμε ήδη δρομολογήσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη φάση για εμάς ήταν ε, η φάση διαβούλευσης με διαφόρους διαφορεμένους φορείς σε συνεργασία με την Επίτροπο Γιούροβα οργανώσαμε ακριβώς πριν ένα έτος, δηλαδή τον Απρίλιο του 2016, ένα συνεργατικό, μια συνεργατική εκδήλωση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό, αυτή η εκδήλωση. Συμμετείχαν πολύ ενδιαφερόμενοι από ένα ευρύ φάσμα, κάλυπταν όλους τους τομείς ε, των μεταφορών. Είχαμε τις κυρίες Ταπαρντέλα για σέντρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με τη σειρά τους ε, είχαν ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις και αυτό, αυτή την εκδήλωση εντοπίσαμε κάποιες δράσεις προτεραιότητα. Είχαμε στη συνέχεια ένα ερωτηματολόγιο, το απευθύναμε στα κράτη-μέλη, ε, στις αντιπροσωπευτικέ οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, για να δούμε ποιε δράσει πρέπει να αναλάβουμε, τι, τι μας συστήνουν και η κυρία Μπούλτ επίσης ε, παρουσίασε στο Συμβούλιο Μεταφορών το θέμα το Δεκέμβριο του 2016. Από αυτή τη φάση λοιπόν, την προτεκτική φάση διαβούλευση. Ε, ανεδίσαν συγκεκριμένοι στόχοι για την πρόθεση της ε, γενικής απασχόλησης και τη ισότητας ανδρών γυναικών στον τομέα των μεταφορών. Συγκεκριμένα δύο είναι οι βασικοί άξονες δράσης. Ο πρώτος είναι να προσελκύσουμε περισσότερες γυναίκες στον τομέα των μεταφορών, που αυτή τη στιγμή πλήττεται από ένα έλλειμμα ε, εικόνα, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Ε, εξελίσσονται οι μεταφορές, έχουμε την αυτοματοποίηση, την ψηφιοποίηση, Η πρόσβαση λοιπόν των γυναικών είναι πολύ πιο εύκολη στον τομέα των μεταφορών και των σκηνών σε σχέση με το παρελθόν. Ουσιαστικά εδώ πρέπει να ε, επικοινωνήσουμε για την ε, κατάρρυψη κάποιων στερεοτύπων. Έχουμε δύο βασικά έργα. Το πρώτο είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ελκυστικότητα τα των μεταφορών και έχουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αφορά συγκεκριμένα τις γυναίκες αυτό το έργο, αλλά ε, τα τμήματα της κοινωνίας ε, που θεωρούμε ότι είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν ε, την ε, έλλειψη εργατικού δυναμικού. Μιλούμε δηλαδή για νέους αλλά και για τους νέους και για τις γυναίκες. Θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Είναι σε εξέλιξη αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και φυσικά θα σας διαβιβάσουμε τα αποτελέσματα. Η δεύτερη δράση είναι μια μελέτη επιχειρήσεων, ένα business case για περισσότερη συμμετοχή των γυναικών στις μεταφορές. Εδώ έχουμε στόχο κυρίως τους εργοδότες. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα που είναι πολύ δεδομένα μεταξύ των εργοδοτών, των οποίων πολλοί θεωρούν ότι θα στοιχήσει πιο πολύ στι επιχειρήσει ε, το να προσλάβουν γυναίκε και εμεί θέλουμε να καταδείξουμε το αντίθετο. Δηλαδή, η γυναική απασχόληση είναι ατού, είναι πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Δεν θέλουμε όμως μόνο να προσελκύσουμε περισσότερες γυναίκες στον τομέα του αλλά και να διατηρηθούν ε, οι γυναίκες, να παραμείνουν σε αυτή τη θέση. Δεν θέλουμε να προσφέρουμε ένα ε, φιλικό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό είναι, αυτός είναι ο άλλος άξονας ε, της δράσης μας και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε σε συνεργασία ενεργό συμμετοχή και της ΕΟΚΕ μια πλατφόρμα για την αλλαγή για τους φορείς των μεταφορών η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτούν να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων στο δικό τους επίπεδο. Άρα εδώ στόχος είναι οι επιχειρήσεις, ε, ε, ο κόσμος της εργασίας. Μια πλατφόρμα προσανατολισμένη στη δράση, δεν είναι μια πλατφόρμα συζήτησης. Θα ξεκινήσουμε σύντομα τις εργασίες. Η ΕΟΚΕ Πρέπει να σας πω ότι προετοιμάζει αυτή τη στιγμή μια διερευνητική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό που αναμένεται να εγκριθεί στα τέλη του μήνα. Θέλουμε να την δρομολογήσουμε την πλατφόρμα για την αλλαγή, αυτή την πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, να έχει γίνει αυτό, για να περάσουμε στην επιχειρησιακή φάση. Συμπερασματικά ελπίζω ότι σας έπεισα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει ξεκινήσει συγκεκριμένες, πραγματικά συγκεκριμένες δράσεις ε, για να προωθήσει την γενική απασχόληση και την ε, ισότητα ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων. Θέλω να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία τη σημερινή μερίδα και ελπίζω να μπορέσουμε να βαθύνουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Βεργό και χωρίς καθυστερήσεις ο λόγος στην πρέσβειρά μας. Πρέσβη ή πρέσβυρα προτιμάτε. Πρέσβυρα. Πρέσβη μάλλον. Η κυρία Άζα Βέμπερ. Μόνιμη πρόσωπο της Σουηδίας παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε για την πρόσκληση να έρθω να σας απευθυνθώ και που διοργανώσατε αυτό το αυτή την εκδήλωση. Πολύ σωστά προβάλλεται αυτό το θέμα και ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους υπόλοιπους βουλευτές που την σημαντική αυτή συζήτηση τη διατηρούν ζωντανή. Είναι σημαντική εκδήλωση. Και να επενέσω και την Επιτροπή για την πολύ καλή της δουλειά και την Επίτροπο Μπούλτ που έχει οργανώσει σχετικές εκδηλώσεις. Και μία αρκετά πραγματιστική προσέγγιση για το τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα ώστε να εκμεταλλευτούμε το ε, κρυφό του δυναμικό και να αξιοποιήσουμε μια διάσταση που θα, είναι, θα έχει μεγάλο όφελος για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, δηλαδή η ισότητα των φύλων επανέλθει στη σωστή ισορροπία. Όπω είπε και ο συγκεκριτή ο κ. Νίλσον, χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει επίγνωση του τι δείχνουν τα στοιχεία και οι αριθμοί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενημερωμένοι. Γι' αυτό τη σύντομη παρουσίασή μου θα τη διαιρέσω σε δύο τμήματα. Ένα γενικότερο για την ισότητα των φύλων και πώ το αντιμετωπίζουν αυτό στην Σουηδική κυβέρνηση και ένα που θα ασχολείται ειδικότερα με το θέμα των μεταφορών και πώ το επεξεργαζόμαστε. Γενικά νομίζω ότι είναι θέμα ηγεσία, θέμα επίγνωση των πολιτικών ηθινόντων. Εμεί είμαστε πολιτικοί ηθινόντε ε, στην Ένωση. Αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Το ίδιο και οι κυβερνήσει μα που πρέπει να γνωρίζουν και να ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και αριθμητικών δεδομένων. Εγώ εκπροσωπώ την Σουηδική κυβέρνηση που είναι μια κυβέρνηση φεμινιστική. Θα το δείτε και στη διαφάνεια και θα τις διατρέξω γρήγορα τις διαφάνειες για να δείτε ότι έτσι δουλεύουμε στη Σουηδία, στη Σουηδική κυβέρνηση. Είναι ίση αριθμή ανδρών και γυναικών στην κυβέρνηση Προωθούμε το gender mainstreaming, την ευθυγράμμιση της διάστασης του φύλου, μέσω της ε, συμπερίληψης του σχεδιασμού του προπολογισμού, που είναι ένα βασικό εργαλείο, και όλων των υπόλοιπων δράσεών μας. Δηλαδή, οι προτεραιότητες και οι αποφάσεις μας πρέπει στόχο να έχουν να αυξήσουν την ισότητα των φύλων. Και αυτό μπορεί να γίνεται συστηματικά. Όπως ε, κάθε μέρα τρώμε πρωινό και γεύμα η πολιτική πρέπει να έχει επιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο στους ανθρώπους και τις, στους άντρες και τις γυναίκες που είναι όλοι άνθρωποι. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το θέμα. Η ενημέρωση, η γνώση είναι κάτι το διαρκές και θα πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει επίγνωση, όπως και η Επίτροπος Μπούλτ έχει ε, εντοπίσει, προωθώντας όλα αυτά τα ζητήματα στη χάραξη πολιτικής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξισορρόπηση των φύλων και τις γενικότερες προοπτικές. Σκοπός είναι οι άντρες και οι γυναίκες να έχουν την ίδια εξουσία να διαμορφώνουν την κοινωνία και τη ζωή τους. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει αναγκαστικά αυτή τη στιγμή και αυτός χρειάζονται συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι για να προωθηθεί αυτός ο σκοπός και τα σημεία που αναφέρονται εκεί είναι πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να είμαστε σε θέση να έχουμε την ίδια προσέγγιση προς τους άνδρες και τις γυναίκες στον τομέα των μεταφορών λόγου χάρη, αλλά και σε όλους τους τομείς. Η ισότητα των φιλών αφορά τα τρία ρο. Την εκπροσώπηση, την, ε, τα δικαιώματα και γι' αυτό θα πρέπει να χτίσουμε τις, ε, να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για τη γονική άδεια και ούτω καθεξής. Είναι προϋποθέσεις ώστε άνδρες και γυναίκες να μπορούν να, να είναι πλήρη μέλη της κοινωνίας και να εργάζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους τομείς όπως των μεταφορών. Έχουμε μια προτεραιότητα για τα θέματα αυτά εδώ και πολύ καιρό και μεταμορφώνει όλη τη χάραξη πολιτικής. Από καιρό το ίδιο και για τις κρατικές εταιρείες και οργανισμούς. Και εκεί ε, χρειάζεται να υπάρξει αυτή η διάσταση με κάποια πρότυπα. Στον τομέα των μεταφορών έχουμε μόνο 3% ε, μηχανοδηγών λόγου χάρη στους σιδηροδρόμους. Δεν είναι καλός αριθμός, δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο χαμηλός αυτός ο αριθμός. Εφόσον το κράτο λοιπόν έχει στην ιδιοκτησία του εταιρείε και υπάρχουν και επικεφαλεί αυτών των επιχειρήσεων, θα πρέπει να φροντίσουμε η διάσταση των φύλων να ενσωματωθεί. Ε, υπάρχει ε, πρόταση για τη συμπερίληψη τη σωστή ποσόστοση στην νομοθεσία μα και εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Να έρθω τώρα σε πιο ειδικά θέματα που αφορούν ε, την πολιτική των μεταφορών θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ως πολιτικοί ηθήνοντες έχουμε τους σωστούς στόχους για να βελτιώσουμε το γενικότερο τοπίο και να καταλήξουμε να έχουμε καλύτερη και πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση της παρουσίας των γυναικών, πιο εξισορροπημένη εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα των μεταφορών και γενικότερα στην παρουσία τους σε θέσεις κλειδιά ώστε να αποτελέσουν και πρότυπο. Για να το κάνουμε αυτό έχουμε ένα λειτουργικό στόχο, την προσβασιμότητα, και έχουμε και ένα στόχο πιο θεωρητικό, ασφάλεια, περιβάλλον και υγεία. Και οι δύο αυτοί στόχοι σκοπό έχουν να βελτιώσουν την διάσταση της ισότητας των φύλων. Ο κλάδος των μεταφορών χρειάζεται άντρες και γυναίκες να βρίσκονται και να εμπλέκονται ε, με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, άντρες και γυναίκες μετακινούνται με διαφορετικούς τρόπους χρησιμοποιούν τον τομέα των μεταφορών διαφορετικά. Αλλά ως πολιτικοί θυνούντες πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη και οι επιλογές μας να είναι τεκμηριωμένες. Να ξέρουμε γιατί διαλέγουμε τι και τι προϋποθέσεις απαιτούνται. Ώστε να υπάρχει μια εξισορροπημένη εκπροσώπηση των φίλων στον τομέα των μεταφορών. Για να γίνουν αυτές οι σωστές επιλογές... Έχουμε την Eurostat για παράδειγμα. Το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ξέρουμε και εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία για να δούμε τι διαφορέ υπάρχουν. Εάν οι άντρε και οι γυναίκε χρησιμοποιούν τι ε, δημόσιε κοινωνίε με τον ίδιο τρόπο, εάν χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά του διαφορετικά, εάν ε, κάνουν διαδρομέ μεγάλη διάρκεια. Υπάρχουν διαφορέ και μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικέ νομοθετικέ επιλογέ. Γι' αυτό Πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία ετησίω και να μελετώνται και για τι ταξιδιωτικέ συνήθειε και για τι ε, επαναλαμβανόμενε συμπεριφορέ, ε, τι ευκαιρίε στην αγορά, τη χρήση των ε, οχημάτων, την ασφάλεια. και για το μερίδιο, για το ποσοστό ανδρών και γυναικών σε διοικητικά συμβούλια και γιατικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις. Χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες και γι' αυτό έχω παραθέσει και μερικές γραφικές παραστάσεις για το πώς έχουν ε, διοργανωθεί όλα αυτά, για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν διαφορετικά τις μεταφορές. Οι άντρες κάνουν περισσότερες διαδρομές για τη δουλειά τους. Οι άντρες και οι γυναίκες παίρνουν περίπου τον ίδιο χρόνο ταξιδεύοντας. Τα βλέπετε. Να τα. Οι άντρες όμως οδηγούν περισσότερο με τα αυτοκίνητα από ότι οι γυναίκες. Είναι κάποια βασικά στοιχεία, αλλά ε, επηρεάζουν και τη θεώρησή μας του συστήματος μεταφορών για να ξέρουμε πώς το χρησιμοποιούν ακριβώς οι χρήστες. Οι συνήθειες και οι συμπεριφορές διαφέρουν. Έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε και ένα γενικότερο πλαίσιο για το πόσο ελκυστικό είναι αυτό ο τομέα και να εντάξουμε και τι κατάλληλε ευκαιρίε για άντρε και γυναίκε. Υπάρχουν και βασικά οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με όλο αυτό και με τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Θα μπορούσε κανεί να τα μελετήσει μόνο και μόνο από οικονομική σκοπιά για να λάβει υπόψη τη διάσταση τη ισότητα των φύλων. Επί της ουσίας δηλαδή πιστεύουμε ότι το να επιδιώξει κανείς αυτούς τους στόχους και να αναγκάσει τον εαυτό του πολιτικό να ασχοληθεί περισσότερο με τους αριθμού και τα στοιχεία, την κατάσταση που ανέφερα προηγουμένω, τα, στατιστικά στοιχεία, αυτό μας κάνει να γνωρίζουμε καλύτερα και να προετοιμαζόμαστε καλύτερα για να προσδώσουμε τα σωστά κίνητρα ω πολιτικοί ευθύνοντες και οι άντρε και οι γυναίκε να μπορούν να χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο το σύστημα μεταφορών, το δίκτυο μεταφορών και να αξιοποιούν τι ευκαιρίε που προσφέρει στι θέσει εργασία. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για το μέλλον. Να είμαστε έβδομοι έχουμε ίση εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά τι θέσει εργασία των τομέα μεταφορών. Είναι ένα δυναμικό που δεν το έχουμε καταληφθεί ακόμη και πρέπει να το αντλήσουμε. Ανυπομονώ για τη συνεργασία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και για αυτό τον κατάλογο επιτρεπτήτων και βεβαίω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλου του Ευρωβουλευτέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέμπερ, για την εξαντλητική σας παρουσίαση, όσο και κατατοπιστική, ε, θα επανέλθω συνέχεια σε όλα αυτά τα θέματα που μας αναφέρατε. Ακολουθεί η κυρία Τίλινγκ, πολιτική γραμματέα των οδικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις οδικές μεταφορές. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που καλέσατε τα συνδικάτα να εκφράσουν την άποψή τους σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που συνδέεται με το μέλλον των μεταφορών και την αγορά εργασία σε όλους τους κλάδους των μεταφορών. Είδαμε κάποια σχετικά στοιχεία αριθμητικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δικά μας συνδικάτο ε, λέγει ότι η προσέλκυση γυναικών στις μεταφορές δεν έχει να κάνει μόνο με το image και τα στερεότυπα ε, και τα κλισέ. Η εικόνα που δίνεται όμως δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Στην Ευρώπη σήμερα ο κόσμος ε, περιμένει ε, συγκεκριμένα πράγματα από την εργασία του και περιμένει να έχει και χρόνο για την ιδιωτική ζωή. Όταν είναι θέματα λοιπόν γυναικών στις μεταφορές, το είδαμε και στην Επιτροπή Γυναικών στην εποχή του κομμουνιστικού μπλοκ, και ζητώ συγγνώμη ε, που είμαι κάπως μαχητική και, και αντιφατική, είχαμε πολύ περισσότερες γυναίκες οδηγούς ε, φορτηγών ή οδηγούς τραμ. Τότε, ε, όταν αποφύτησα ήταν προγραμματισμένη η οικονομία, δεν είχαμε επιλογή. Μας είπαν, μου εσύ θα γίνεις οδηγός φορτηγού ανεξαρτήτως ε, προέλευσης, καταγωγής κτλ. Σήμερα έχουν ευκαιρίες και επιλογές ε, τα κορίτσια και οι γυναίκες και θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές και να εφαρμοστούν και στον κλάδο των μεταφορών, σε όλες τις μεταφορές, όλα τα μέσα μεταφοράς, για να ε, προσελκύουμε και να διατηρούμε γυναίκες σε αυτή την απασχόληση. Επανέρχομαι στο θέμα της ποιότητας εργασίας και της ποιότητας ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για γυναίκες εργαζόμενες στις μεταφορές, οι γυναίκες που το σκέφτονται. Είναι η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής. Υπάρχει σήμερα ισότητα στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Αυτό συζητείτε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε ισότητα στο σπίτι. Μεγάλο ερώτημα. Οι απαντήσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το ποιος θα απαντήσει από τους παρόντες, αλλά από τη σκοπιά των γυναικών που εργάζονται στις μεταφορές δεν υπάρχει ισότητα στο σπίτι και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ισορροπία δουλειάς και ε, οικογένειας. Ε, στις μεταφορές δεν ε, είναι όλες οι γυναίκες οδηγοί. Δεν μετακινούνται όλες οι γυναίκες. Είναι πολύ λιγότερες εκείνες που μετακινούνται και περισσότερες είναι σε θέσεις γραφείου. Ε, λόγω της οργάνωσης της ε, δουλειά περιμένοντας να μπούμε για την ακρόαση, είχαμε μια συζήτηση μεταξύ μας με κάποιους εκπροσώπους μεταφορικών εταιριών. Και εδώ μιλώ για πούλμαν, ε, για λεωφορεία. Πώς το ερμηνεύουν λοιπόν οι εταιρείε αυτό. Γιατί δεν επιλέγουν να οδηγεί λεωφορείων γυναίκες. Διότι οι ώρες αιχμής που χρειάζεται ένα λεωφορείο είναι οι ώρε που θα πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν τα παιδιά του στα σχολεία, ε, στον παιδικό σταθμό ή να τα φέρνουν στο σπίτι από τον παιδικό σταθμό. 18 λοιπόν, 20% των οδηγών λεωφορείων είναι γυναίκες μόνο. Άρα, τι θα πρέπει να γίνει εδώ. Η Ομοσπονδία μας Πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενη εάν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια φωτογράφηση ε, ε, των καταστάσεων που επικρατούν στις διάφορες μεταφορές στα λιμάνια και σε δύσκολους χώρους και όχι μόνο στο σιδηρόδρομο ή στις αστικές συγκοινωνίες, στα δημόσια μέσα μεταφοράς όπου υπάρχουν περισσότερες γυναίκες. Ε, λοιπόν, το θέμα δεν είναι η στις αστικες κοινωνιε στα δημοσια μεσα μεταφορας οπου υπαρχουν περισσοτερες γυναικες ε, λοιπον το θεμα δεν ειναι η σωματικη κατασταση και η δύναμη των γυναικών, αλλά είναι το αν μετακινούνται ή όχι. Αν είναι σταθερές θέσεις εργασίας σε ένα τόπο εργασίας, σε ένα μετακινούμενο. Ε, λοιπόν, η οχι αν ειναι σταθερες θεσεις εργασιας σε ενα τοπο εργασιας ειναι ενα ε λοιπον η ισοτητα στο σπίτι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί επηρεάζει ε, την ισορροπία εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Επίσης, άλλα θέματα που μας απασχολούν εργονομικά, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, ε, στις μεταφορές που είναι προσανατολισμένες ακόμα στους άνδρες. Και ένα τελευταίο, ένα τμήμα όλων αυτών είναι ε, η βία στο χώρο εργασίας. Από τον Νοέμβριο έχουμε κάνει μια έρευνα μεταξύ των μελών μας για τη βία που υφίστανται οι γυναίκες, παρενόχληση από συναδέλφους ή από τρίτους. 1.350 απαντήσεις πήραμε για να έχουμε κάποιες στατιστικές αλλά και κάποιες μαρτυρίες. Και τι λέγουν οι μαρτυρίες είναι πράγματα που δεν έχουν θέση στο σημερινό κόσμο, ούτε στη σημερινή Ευρώπη. Έχετε γυναίκες οδηγούς λεωφορείων, ας πούμε, ή ε, προσωπικό εξυπηρέτηση εδάφους στα αεροδρόμια, που υφίστανται απίστευτα πράγματα. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύσουμε και ε, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ισχυρές συστάσεις διότι δεν μπορείς να πας σε μια εταιρεία και να την αναγκάσεις να κάνει το α, το β και το γ, αλλά να αποκαλύψουμε την κατάσταση πάντα βοηθάει. Και πάντα έχει επίπτωση αυτό. Να έχει λοιπόν έντονες συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα της θέσης εργασίας. Η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ε, εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε κοινωνικούς εταίρους στις συνδρομικές μεταφορές και στις αστικές συγκοινωνίες που έχουν κάνει δύο έργα. Ο καθένας ε, την τελευταία πενταετία για την ανάλυση, για την καταγραφή της κατάστασης. Τα ίδια αντίστοιχα ισχύουν στην αυτιλία. Έχουμε μια εργαλειοθήκη για την ε, καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης εμπλό και πρέπει εδώ να σας πω ότι οι γυναίκες δεν παραδέχονται δεν αναγνωρίζουν ε, όλες τις καταστάσεις ως παρενόχληση, ως βία. Και αυτό σημαίνει ότι ανέχονται τις καταστάσεις αυτές. Οι εταιρείε λέγουν στου εργαζομένου μεταφορέ και στι γυναίκε ότι κοιτάξτε, είναι τμήμα τη δουλειά σου και κανόνισε να το αντιμετωπίσει. Κάναμε λοιπόν αυτή την έρευνα και αυτό πραγματικά άνοιξε τα μάτια των εργαζομένων στον κλάδο των γυναικών. Ε, και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε πιο έντονη αντίδραση, πιο ε, στιβαρό πυλώνα για την ισότητα των φύλων στην εργασία και τα θέματα που άπτονται ε, των γυναικών. Παραμένω σε πολύ γενικά σχόλια. Ένα τελευταίο. 3% των γυναικών που οδηγούν τραμ μάλλον των οδηγών τραμ στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Αναφέρομαι στη χώρα μου. Η επένδυση στο σιδηρόδρομο στα, μέσα σταθερής ε, τροχιάς είναι πολύ μικρή. Ε, ε αυξάνονται οι ε, αποστάσεις γιατί ο κόσμος ζει στην περιφέρεια και μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων. Ο αδερφός μου οδηγεί τραμ και δεν έχει χρόνο ξεκούρασης ε, στη βάρδια του ουσιαστικά. Φανταστείτε οι γυναίκες. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα εδώ. Θα πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε ο και κλάδο των μεταφορών να είναι ελκυστικός για γυναίκες και να γίνουν πολλές αλλαγές έτσι ώστε να προσελκύονται και να παραμένουν σε αυτή τη δουλειά οι γυναίκες. Ελπίζω να έχουμε επικοδομητικό διάλογο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο στο μέλλον για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup pour... Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Και τώρα το λόγο έχει η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρία Χακστάινερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Μεταφορών που κάλεσε την EBU στην ακρόαση αυτή. Να σας παρουσιάσω συντομία την οργάνωσή μας. Είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση εσωτερικής σε νέα ευρωπαϊκές χώρες ε, προσωπούνται, αλλά και χώρες εκτός Ένωσης. Κάποια βασικά στοιχεία. Η εσωτερική ναυσιπλοεία έχει την επίδοση των 140 δισεκατομμύρια τόνων ε, ανά χιλιόμετρο 515 εκατομμύρια τόνοι δηλαδή εμπορευμάτων, που ουσιαστικά εκπροσωπεί το 7% μόνο του συνολικού των συνολικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, σε χώρε όπω είναι η Ολλανδία, το ποσοστό αυτό είναι πολύ ψηλότερο, 40% για παράδειγμα. Επίση, είναι ένα τρόπο μεταφορά ε, στον οποίο απασχολούνται πάνω από 42.000 άτομα πάνω στα πλοία, εκ των οποίων 30.000 περίπου είναι κινητοί εργαζόμενοι, όπως ε, αναφέρεται αυτό ο όρος στις ε, συμβάσεις εργασίας και 11.000 περίπου αυτοαπασχολούμενοι. Για να σας εξηγήσω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, ζουν πάνω ε, και ταξιδεύουν πάνω σε αυτά τα ποταμόπλια. Και πολλές φορές αυτά, αυτές οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, η γυναίκα και ο άνδρας δηλαδή, και δεν έχουν ακριβώς την ίδια, τα ίδια προσόντα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει γενικότερα τον κλάδο είναι οικονομία κλίμακας, ψηλό ασφάλειας, ε, σχέση κόστος-οφέλους, χαμηλό εξωτερικό κόστος και ε, έλλειψη συμφορήσεων. Έρχομαι στις γυναίκες, στις μεταφορές, που είναι και το θέμα μας. Πραγματικά είναι πρόκληση και στο δικό μας τον κλάδο. Έχουμε αναλάβει εδώ και δύο χρόνια περίπου να διαπραγματευόμεθα με το ETF. Χαίρομαι γιατί είναι και συνάλφος εδώ από το ETF. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν πριν από κάνα δύο-τρία χρόνια και πετύχαμε να έχουμε την πρώτη σύμβαση ε, χρόνο εργασίας όπου ε, αναφέρονταν οι προϋποθέσεις για τους κινητούς εργαζόμενους ε, πάνω στα πλοία. Υπήρχαν γενικά κριτήρια ε, για το χρόνο εργασία ε, που έπρεπε να εκπληρώνονταν, αλλά μάλλον υπόψη και ιδιαιτερότητε του τομέα. Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, συζητούμε επίση ε, και τα ζητήματα στελέχωσης, του, τα πληρώματα. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό στις διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους μας από τις μεταφορές. Πολύ πρόσφατα Είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση να εργαστούμε για τα επαγγελματικά προσόντα, τι επαγγελματικέ δεξιότητε με το ETF. Ξεκινήσαμε με τους καινούς εταίρου ε, μια συνεργασία για να ε, προβούμε στην εναρμόνιση των προσόντων ε, και των κύκλων σπουδών τη εκπαίδευση. με στόχο το επόμενο βήμα που είναι ακριβώς πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη θεωρική ναυσιπλοεία. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που αυτή τη στιγμή είναι από διαπραγμάτευση. Συμμετέχει και η δική σας επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Χαρακτηριστικό είναι ένα νέο σύστημα εκπαίδευση που θα βασίζεται στις ε, επιδόσεις και όχι μόνο στην πρακτική όχι μόνο στην πράξη. Ένα από τα βασικά κριτήρια είναι ότι στόχο έχει να βελτιώσει την κινητικότητα καλά εκπαιδευμένων εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπα και οι προλαλήσαντες, οι προλαλήσασες κυρίως ότι στον τομέα των μεταφορών γενικά, αλλά και στην εσωτερική ναυσικλία συγκεκριμένα, αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη ε, ελκυστικότητα, να ε, ενισχυθεί εικόνα, να μπορεί να προσελκύσει ο κλάδος περισσότερους εργαζομένους. Αυτό ξεκινάει από την ε, βάση, από τα σχολεία. Θέλουμε να μπει ε, στη διδακτέα ύλη, στο πρόγραμμα σπουδών και μάλιστα από νωρί, από μικρή ηλικία, πριν αποφασίσει ένα νέο ε, τι επάγγελμα θα ακολουθήσει, να δημιουργήσουμε ευαισθητοποίηση απέναντι στι διάφορες του διάφορου τρόπου μεταφορά στην περίπτωσή μα για την εσωτερική ναυσιπλοεία, θέλουμε να προσελκύσουμε νέου άνδρε και νέε γυναίκε Επίσης, ε, η ιστορική ναυσιπλοεία χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτό θα είναι μια όλο και πιο ε, μεγάλη πρόκληση στο μέλλον. Και στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και στο πλαίσιο αυτής της πρότασης και άλλων προτάσεων, θέλουμε να έχουμε υποστήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Με βάση τα κριτήρια και τι συμφωνίες που έχουμε για το ωράριο εργασία και τι άλλε συμφωνίες. Νομίζουμε ότι έτσι θα καταστεί πιο ελκυστικό ο κλάδος, θα βελτιωθεί η εικόνα του, πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Χρειάζονται περισσότερες γυναίκες, χρειάζονται περισσότεροι νέοι στον κλάδο αυτό. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ. Merci beaucoup για όλες αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Πρέπει να πω ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών διαπιστώνω, ε, γιατί συμμετέχω σε πολλά συνέδρια και ημερίδες ε, των αερομεταφορών, συνδρομικών μεταφορών, οδικών μεταφορών και διαπιστώνω ότι καμιά φορά αισθάνομαι πάρα πολύ μόνη μου στα πάνελ γιατί οι ομιλητές είναι 100% άνδρες και είναι προς τιμή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε δύο γυναίκες και πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών του Κοινοβουλίου και επίτροπο σε ένα κλάδο που ανδροκρατείται. Αλλά το 50% των γυναικών χρησιμοποιούν τις μεταφορές. Et ça, ça va être un des défis du 21e siècle, mais que ces effectifs, on les retrouve. Και αυτό είναι μια πρόκληση του 21ου αιώνα. Και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη τους οι εταιρείε όταν παίρνουν τις αποφάσεις τους. Και θα πρέπει να υπάρχει παρουσία γυναικών και στους θεσμούς και πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να έχουν περισσότερες γυναίκες και σε άλλα επαγγέλματα που θεωρούν το ανδρικά ε, στο παρελθόν με συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν θα πρέπει να παραμελούμε ε, το γεγονός ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση πάντα εκ των προτέρων. Δηλαδή από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, για να μπορούμε να προσανατολίζουμε τα κορίτσια. Γιατί όταν έχουμε επαγγέλματα όπως πιο των θετικών επιστημών, των τεχνικών ε, επαγγελμάτων, θεωρούν οι γυναίκες ότι δεν είναι για μας αυτές οι δουλειές. Όχι. Να ανοίξουμε τις πόρτες και να δείξουμε ότι και οι γυναίκες είναι εξίσου υπεύθυνε. Θα πρέπει από νωρίς να αρχίζει αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός από το σχολείο ότι κοιτάξτε να δείτε και για εσάς τα κορίτσια είναι αυτές οι εταιρείε. Αυτή ήταν η μικρή πολεμική μου ή αρχή. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους και θα αρχίσουμε από τον κύριο Μπαχ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να διαπιστώσω ότι το σύνολο του κλάδου των μεταφορών δεν χαίρει της καλύτερης δυνατής εκτίμησης. Δεν έχουμε απλώς ε, λίγες γυναίκες οδηγούς, αλλά γενικότερα ε, έχουμε έλλειψη οδηγών. Και αυτό ε, το βλέπουμε και να επιμερίζεται στους διάφορους κλάδους. Κυρία Πρόεδρε, είπατε κάτι προηγουμένως σύντομα στην παρέμβασή σας ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες που να ενδιαφέρονται πολύ για τα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα, τεχνικό κλάδο. Ισχύει αυτό. Και το υπογραμμίζω και το υποστηρίζω αυτό που λέτε. Και θα μπορούσαν, φαντάζομαι, να συμφωνήσουν και τα μέλη του πάνελ. Βλέπουμε τώρα τις νέες ευκαιρίες και τις νέες εξελίξεις, μεταφορές με ψηφιοποίηση, με αυτοματοποίηση κτλ. Άρα θα μας λείψουν ακόμα περισσότερες ε, δεξιότητες και εργαζόμενοι. Αν δούμε τι γίνεται τώρα ε, στα πανεπιστήμια και στις τεχνικές σχολές, ε, είναι περίπου 100% άνδρες οι φοιτητές εκεί. Λοιπόν, για το θέμα της ε, ισορροπίας και του συνδυασμού εργασίας με την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή ζωή, παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για να εργαστούν οι γυναίκες στις μεταφορές. Το είπε και η κυρία Τίλινγκ, ότι έχει διαπιστώσει ξεκαθαρά ότι αν κοιτάξετε τι είναι οδηγή λεωφορείων στις αστικές συγκοινωνίες ή ε, μεταφορές, αστικές συγκοινωνίες, έχουμε γυναίκες οδηγούς, αλλά όταν πρόκειται για ε, εταιρείε ε, λεωφορείων με πούλμα που κάνουν μακριά ταξίδια στο εξωτερικό, εκδρομές κτλ. Είναι δύσκολο να δεις γυναίκες οδηγούς, είναι περισσότεροι άνδρες. Εδώ χρειάζεται ε, μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορεί μια γυναίκα να συνδυάζει την εργασία της με την οικογένειά της, ακόμα και αν έχουν γίνει πολλές πρόοδοι. με τις διάφορες μορφές ε, διακοπών και ταξιδιών και αδειών. Ε, αυτό παραμένει πρόβλημα και υπάρχει χάσμα όχι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και μεταξύ των διαφόρων κρατών. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπερκό αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε. το οποίο θέλει να αναβαθμίσει και την εικόνα που δίνουν οι μεταφορές θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Έχετε κάποια πρώτα στοιχεία ήδη. Και αν ναι, θα μπορούσατε να μας τα διαβιβάσετε. Να μας δώσετε μια γεύση. Γενικά. Πραγματικά θέλω να σας εκφράσω την εκτίμηση και την αναγνώριση μου. Έχετε κατανοήσει τα προβλήματα, τα έχετε εντοπίσει τα προβλήματα, οι λύσεις μας λείπουν ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παχ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και συγχαρητήρια γιατί επιτέλους καταφέραμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση γιατί θυμάστε ότι είχαμε ένα σεμινάριο ε, με τις κυρίες Γιούροβα Μπούλτς είχαμε ζητήσει πολλές φορές ε, να οργανωθεί αυτή η Τέλος πάντων. παρόλα αυτά λυπούμε για τρία πράγματα. Πρώτον που δεν ήρθε η Επίτροπος. Στη Σκοτία θα είναι μάλλον. Έτσι φαίνεται από το Twitter στο οποίο επιδίδεται με μεγάλο ζήλο Πρέπει να είναι στη αλλά τέλος πάντων. Θα ήταν καλό να είναι εδώ. Το δεύτερο. Ο τίτλος είναι λίγο αξιοθρύνητος για το όλο μεταξύ μας. Μιλάμε για τις γυναίκες. Οι γυναίκες θα λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης σπόρων και μετά Έχουμε τους ετούντες άσυλο και πρόσφυγες που θα λύσουν τα υπόλοιπα προβλήματα. Εντάξει τώρα, σοβαρευτούμε. Το θέμα γιατί υπάρχουν τόσο λίγες γυναίκες στον τομέα των μεταφορών και στο τιμόνι όσο οδηγείται ε, στις φορτηγίδες είτε στα τρένα είτε οτιδήποτε και γιατί είναι τόσο λίγες οι γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια και στι δημόσιε επιχειρήσει, που έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτική ποσόστοση πόσο είναι δημόσιε επιχειρήσει, όπω ανέφερε και η πρέσβη, ε, και έτσι θα είχαμε πολύ περισσότερε δυνατότητε. Θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε να συμμετέχουν περισσότερε γυναίκε. γιατί έχουν ε, ιδιαίτερες γνώσεις και η χρήση που κάνουν των μέσων ε, μεταφοράς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό των μεταφόρων. Τέλος, Ενδιαφέρον θα ήταν και το είχαμε πει ίσως στο μέλλον θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάτι. Καλό θα ήταν να έχουμε συμμετοχή των γυναικών στον έλεγχο των ε, στην καθοδήγηση. Ε, υπάρχουν, ε, το είχαμε πει, θα έπρεπε να είχαμε γυναίκες ε, πιλότους, ε, γυναίκες οδηγούς φορτηγών, ε, κυβερνήτες φορτηγίδων, να έρθουν εδώ να μας πούν πέντε πράγματα και να ξέρουμε γιατί δεν προσαρμόζονται μεταφορές, όχι στις γυναίκες, γιατί το πρόβλημα για την συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες αλλά γενικότερα και για την κινητικότητα. Έχουμε και τη διελτουργικότητα, είναι ένα θέμα και αυτό. Δεν θα έπρεπε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε τη συμφιλίωση της οικογενειακής ε, και επαγγελματικής ζωής για τους κινητούς εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες στον 21ο αιώνα. Νομίζω δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μια πιο ολιστική προσέγγιση, όχι μια αμυγός μια προσπάθεια αμυγός να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης γυναικών στον τομέα των μεταφορών. Έρχομαι στην Σουηδέζα πρέσβη. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσον έχετε μελέτες και στοιχεία συγκεκριμένα, γιατί θα ήθελα πολύ να γνωρίζω. Έχετε στοιχεία για τις πόλεις μόνο. Υπάρχουν κάποιες μακρές ε, ε, διαδρομές ε, με αστικά λεωφορεία μεταξύ πόλεων. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε στοιχεία και για την νυχτερινή εργασία θα ήθελα να μου πείτε, γιατί και στις δημόσιες συγκοινωνίες αλλά και στις υπόλοιπες ε, και στις ιδιωτικές μεταφορές έχουμε το πρόβλημα με την νυχτερινή εργασία. Είναι και αυτό ένα θέμα αντίληψης. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπεργκό, που τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΟΥΒ πολύ επιτυχημένα χειρίστηκε το πολύπλοκο αυτό ζήτημα. Ενδιαφέροντα αυτά τα project που μας αναφέρατε και το είχαμε ζητήσει και εμείς, γιατί θέλαμε να υπάρξει μια αλλαγή νοτροπίας και εστίασης μεταφορές, αλλά θέλω να ξέρω αν υπάρχει μια ολιστική στρατηγική στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ όχι μόνο στη μονάδα αυτή, αλλά όλη η γάμα δέλτα μου νομίζω θα έπρεπε να ακολουθεί μια ολιστική στρατηγική, όπως έγινε για παράδειγμα με τη γάμα δέλτα έρευνα. Στο σεμινάριο υπήρχε προσωπικό που ήξερε πολύ καλά πώς ό,τι έχει να κάνει με την αντίληψη και τον τρόπο σκέψης μιας γενικής διεύθυνσης όπως η ΓΑΜΑ μπορεί να συμπεριλάβει και θέματα ισότητας. Ε, Μας είπατε για η πρόεδρος. Μπορείτε να ολοκληρώνετε. Ναι, ναι, θα ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυρία που έλεγε για κάτι για τι κομμουνιστικέ χώρε δεν μα προτείνεται, φαντασμένα να γυρίσουμε στο παρελθόν και από τη συνδικαλιστική πλευρά. Προτάσει που κάνετε και τα σχετικά με τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματική ζωή, νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο εμφανή. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ κυρία Γέλα Σέντερ. Λούφιξον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα και το έχω πει επανειλημμένος ότι σε αυτό το τομέα δεν υπάρχουν και πολλές συνάδελφοι γυναίκες, όντως. Σε εθνικό επίπεδο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γυναίκες που θα ήθελαν να δουλέψουν. Όμως Ε, υπήρχαν γυναίκες που ε, πήγαιναν να κάνουν τέτοιε δουλειές γιατί έβγαιναν και χρήματα τότε από αυτές τις δουλειές και χρειάζονταν τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ανταγωνισμό με όλα τα άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται, με το καμποτάζ και με όλες τις άλλε μορφές μεταφοράς. Σε χώρε όπως η Σουηδία οι μισθοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και πρέπει να πω ότι υπάρχει και ένα θέμα ελεύθερης κυκλοφορίας εδώ. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να είναι ε, ξεκάθαρος προς αυτή την αρχή, η οποία θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η κατάσταση στην πραγματικότητα έχει να κάνει με το ότι κάποιο μπορεί να χρειάζεται να περνάει τη μέρα του μέσα σε δύο τετραγωνικά μέτρα ή να μην βρίσκει εύκολα πάρκινγκ και στάθμευση στην καθημερινή του δουλειά. Για παράδειγμα, τα ταξί ή άλλοι οδηγοί μπορεί να έχουν πολύ επιμεκημένα ωράρια εργασία ή να αντιμετωπίζουν απειλές εντός του ταξί, για παράδειγμα. Ίσως θα πρέπει σε ορισμένες ε, περιπτώσεις να δουλεύει κανείς ένα πεντάωρο, εξάωρο, μερικές φορές μπορεί να συμπληρώσει κάποιες βραδινές ώρες δουλειάς. Είναι πολύ δύσκολο να τα συνδυάσει αυτά με την οικογενειακή του ζωή. Και χρειάζονται και κάποιες ώρες ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί αποφασίζουν να πάρουν το αυτοκίνητο, επί παραδείγματι. Προσπαθούμε να εργαστούμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Μεν, όμως κάποιες φορές καταλήγει κανείς να είναι στη γύρα όλη τη μέρα. Υπάρχει μια σειρά από προβλήματα λοιπόν σε ό,τι αφορά τις, ε, τα προσόντα, την ε, κατάρτιση στον τομέα των μεταφορών. Πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ενδιαφέροντα αυτά που ακούω. Ε, να με μια μικρή κριτική. Το είπε και η συνάδελφός μας Αγιάλα Σέντερ. φαίνεται ότι έχουμε μπει σε ένα χάος, ότι και πνιγόμαστε και ξαφνικά σκεφτήκαμε α, γυναίκες να φέρουμε για να καλυφθεί αυτό το κενό και να βελτιωθεί η εικόνα των μεταφορών. Συνδέεται και πάλι η παρουσία των γυναικών με βελτίωση της εικόνας που δίνει ο κλάδος. Λίγο αντιφατικά είναι αυτά με τα όσα ακούμε και με την προοπτική που θα πρέπει να δώσουμε σε αυτό το θέμα. Παρόλο που έχουν αποθετικά πράγματα, λοιπόν, ξεκινώ με μια μικρή ε, κριτική. Ε, όλα αυτά ωραία που μας λέτε, ε, αλλά έχω μια ερώτηση που θα μπορούσε κάποιος να μου απαντήσει, οποιοδήποτε από εσά. Σε άλλες ε, εκθέσεις μιλούμε για την εξέλιξη του κλάδου των μεταφορών με την αυτοματοποίηση κυρίως των συστημάτων μεταφορών. Μιλάμε τώρα πια για drones, για μεταφορές χωρίς οδηγούς. Η Ιαπωνία τι έκανε. Εδώ υπάρχουν φορτηγά που κυκλοφορούν μόνο τους στον αυτοκινητόδρομο στην Ιαπωνία χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Μιλάμε ότι ε, προς τα εκεί ε, εξελίσσεται ο κλάδος και η απασχόληση με όλα τα καμπανάκια που μπορούν να ανάψουν και για τα ρομπότ. Εσείς πώς βλέπετε να διαγράφετε το μέλλον ε, με αυτά τα θέματα που μας απασχολούν στις άλλες εκθέσεις. Στη συνέχεια, αν το 60% των πτυχίων στην Ευρώπη και των πτυχιούχων είναι γυναίκες, πώς θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις γυναίκες σε τέτοιες θέσεις εργασίας που χρειάζονται λιγότερα προσόντα και λιγότερη μόρφωση. Ενώ οι γυναίκες είναι το 60% των πτυχιούχων. Και βλέπουμε να διευρύνεται η ψαλίδα και το χάσμα. Όλο και περισσότερε γυναίκες φοιτούν στα πανεπιστήμια από άνδρες. Και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τέιλορ. Um, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε δεν μου δίνεται και πολύ συχνά δυνατότητα να μιλήσω με όρους, να μιλήσω για ανδροκεντρική ε, προσέγγιση. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση της, ε, μεταφορ... της πολιτικής μεταφορών. Ανδροκεντρική. Η στόχοι ισότητας των φύλων, κοινέ πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την χάνουν λόγω των πολιτικών που ισχύουν σήμερα, που εφαρμόζονται. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον αυτή την έκθεση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μιλάω για την έκθεση που μιλάει για τη φύση των μεταφορών. Ότι οι γυναίκες ε, πιο πολύ κάνουν ταξίδια, ενώ οι άνδρες κάνουν ταξίδια για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η, μετα... η πολιτική μεταφορών ε, σε μεγάλο βαθμό σχεδιάζεται από τους άνδρες και απευθύνεται σε άνδρες. Γι' αυτό τη να χαρακτηρίζω άνδρο κεντρική. Οι γυναίκε φαίνεται ότι πιο πολύ χρησιμοποιούν τι δημόσιε συγκοινωνίε και ε, τα πόδια του. Ενώ οι άνδρε ε, με αυτοκίνητο πιο πολύ ταξιδεύουν. Νομίζουν ότι είναι και σημαντικότερη, το σημαντικότερο της μεταφορών, ιδιωτικές μεταφορές, το αυτοκίνητο. Η ισότητα των ε, φύλων ε, και τα προβλήματα ε, που δημιουργεί επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν άντρες και γυναίκες, τις δυνατότητες κινητικότητας, την ποιότητα επίσης των μεταφορικών υπηρεσιών. Οι γυναίκες και οι άντρες ταξιδεύουν για διαφορετικούς λόγους για την εργασία, για τα ψώνια, κοινωνικές συναναστροφές, ε, ε, επαγγελματικούς σκοπούς κτλ. Αλλά βασίζεται η χάραξη ε, της πολιτικής στις ανάγκες των ανδρών ουσιαστικά. για να φτάσουμε εδώ που, από εδώ που είμαστε, εκεί που πρέπει να φτάσουμε, να, στα στόχους ισότητας των φίλων, θα πρέπει άρδιν να αναθεωρηθεί η πολιτική μεταφορών και γι' αυτό επικροτώ την πολιτική που αναφέρεται στη μελέτη. Θα με ενδιαφέρει για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι, θα ολοκληρώσω. Να δω περισσότερα για αυτό το θέμα της απασχόλησης ε, στις μεταφορές στην Ήπεθρο. 13% εδώ είναι οι γυναίκες μόνο. Και μιλούμε κυρίως για οδικές μεταφορές. Για την Ήπεθρο μιλάω πάντα και νομίζω ότι αυτή είναι μια μείζων πρόκληση. Επίσης θα πρέπει να τονώσουμε, να προωθήσουμε την αλλαγή και η Κομισιόν νομίζω ότι θα πρέπει ενεργά να προωθεί την ισότητα των φύλων σε όλα τα θέματα των μεταφορών. Και στο επικείμενο έργο της να περιλάβει αυτή τη διάσταση. Ολοκληρώνοντας, πριν από ένα χρόνο, πήρα ένα από τα οχήματα ε, του Κοινοβουλίου και η Σοφέρη ήταν γυναίκα και τη ρώτησα πόσες γυναίκες οδηγούς έχουμε στο κοινοβούλιο. Δύο μου είπε, από 100 σοφέρ. Θα έπρεπε να ξέρει αυτή η Επιτροπή ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα λοιπόν. Έχουμε ένα νέο στόλο, Mercedes, Mercedes 220 και Αλφα Ρωμαίο. Έχουμε 100 οδηγού πάντα, αλλά ξέρετε κάτι, ξεκολουθούμε να έχουμε μόνο δύο γυναίκες σοφέρ. Κάτι πρέπει παραπάνω να γίνει για να φτάσουμε την πραγματική ισότητα των φίλων. Εδώ, σε αυτό το μέρος που υποτίθεται ότι είναι και πραγματικός στόχος για τον οποίο και εγώ είμαστε η ισότητα των φίλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο που διοργανώσαμε σήμερα το πρωί αυτή την ακρόαση. Αν κοιτάξετε όμω γύρω σα, δεν θα φανταστείτε ότι είναι μέγα πολιτικό το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα και απογοητευτικό. Όλοι στην Επιτροπή Μεταφορών λένε ωραία λόγια και μεγαλόστομα, αλλά όταν φτάσει η ώρα της αλήθειας, έχουμε δουλειά σε άλλες επιτροπές. Συμφωνώ πάρα πολύ με τον Ζογς Μπαχ. Χρειάζεται να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο οι γυναίκες στις ευρωπαϊκές μεταφορές. Αυτό είναι προφανέστατο. Εγώ έχω πολύ καλές εμπειρίες στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες έχουμε γυναίκε μηχανοδηγούς στο σιδηρόδρομο και αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα στο τρένο. Είναι ε, πιο ήρεμη η ατμόσφαιρα, ε, λιγότερο ε, φαλοκρατική, λιγότερο άνδροκρατούμενη και ε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ταξίδι. Έχουμε λοιπόν έλλειψη προσωπικού και τίθεται το εξή ερώτημα και ρωτώ την κυρία Βέμπερ από τη Σουηδία και την κυρία Τίλινγκ. Τι θέλουμε τώρα, την απόλυτη ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Αυτό με δυσκολεύει εμένα. Ακούσαμε για την νυχτερινή εργασία από την κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευτυχώς έχουμε και παιδιά που πρέπει κάποιος να τα αναθρέψει. Και είναι εύκολο να πείτε ότι ο άντρας θα παίξει τον ίδιο ρόλο, αλλά η ζωή είναι λίγο πιο ρεαλιστική από το να πούμε ότι τα ισοπεδώνουμε όλα ή τους ή, ε, τα όλους. Και έχω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε πιο ε, ασφαλείς σταθμούς στάθμευσης. Δηλαδή, ε, όταν σταματάει σε ένα πάρκινγκ, ε, ένα φορτηγό θα πρέπει να έχει την ευκαιρία ο οδηγός ή η οδηγός ε, με άνεση και με ασφάλεια να πιέσει την τουαλέτα, να κάνει ντους κτλ. Λοιπόν, προσέξτε, ε, στην εσωτερική ναυσιπλοεία οι γυναίκες, οι σύζυγοι των πλειοκτητών ε, είναι ναυτικοί και ίδιες στις εσωτερική ναυσιπλοίες στις φορτηγίδες και μοιράζονται και ώρες ατελείωτες ε, πλέον ε, στα ποτάμια. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση, αλλά μήπως να είμαστε λίγο πιο προσγειωμένοι και να μην ζητάμε το 50-50. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φανταγκάμπη κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ε, εδώ στην ακρόαση βλέπω και το ίδιο και εκτό αίθουσα. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε παίρνουν πολύ σοβαρά το ζήτημα αυτό. Μα ενδιαφέρει ω προ την ισότητα των φύλων και τη διαφοροποίηση ε, αυτό που βλέπουμε να ε, υπολογίζεται γενικότερα για την αγορά εργασία ότι μέχρι το 2050 μπορεί να έχουμε πετύχει πραγματική ισότητα σε όλα τα εργασιακά και στον κλάδο των μεταφορών θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό καλωσορίζω όλε τι παρουσιάσει που έγιναν σε σχέση με αυτό. Καταγράφω αυτά που μα είπε η Επιτροπή για την ε, Γενική Διεύθυνση για που ασχολείται με τα θέματα αυτά και την ευθυγράμμιση τη διάσταση τη ισότητα των φύλων. Αλλά πρέπει να δούμε πού θέλουμε να πάμε, διότι ο κλάδο των μεταφορών βρίσκεται τις τελευταίες προτεραιότητες ε, της εργασιακής ποιότητας και αυτό συνδυάζεται και με όσα ακούστηκαν για τον αντίκτυπο στις γυναίκες και όλος ιδιαιτέρως ε, ε, στο εργασιακό δυναμικό των μεταφορών σε όλους τους κλάδους. Εάν δούμε την ε, βασική έρευνα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εργασιακές συνθήκες, κάθε μέτρο που αφορά την ποιότητα της εργασίας έχει τελευταίο τον κλάδο των μεταφορών, δηλαδή βρισκόμαστε στον πάτο του πάτου. Εδώ λοιπόν ε, τα, ε, τα διαλύματα για την ανάπαυση, τα υποχρεωτικά διαλύματα, δεν είναι ότι δεν υπάρχει ότι δεν για τους άντρες, αλλά οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες για τις γυναίκες. Και το πώ διοργανώνονται οι θέσει αυτέ εργασία έχουν να κάνουν με το κατά πόσο οι γυναίκε παίρνουν αυτέ τι δουλειέ. Και γενικώ για την Επιτροπή μα, ε, κάτι που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω. Πρόοδο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα. Πού είναι αυτή, πού είναι για τι καλέ θέσει εργασία. Κάποια από αυτή την πρόοδο θα πρέπει να είναι νομοθετική και όχι απλώ εθελοντική. Γι' αυτό λοιπόν που είπε ο κύριο Μπαχ, πού είναι οι λύσει, τι θα κάνουμε για όλα αυτά στον τομέα των μεταφορών, όλο ιδιαίτερω. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και ιδίω σε ό,τι αφορά τι ευκαιρίε που θα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να υπάρχουν ε, ε, διαφοροποιημένε συμβάσει και διαφοροποιημένη πρόβλεψη στι δημόσιε προμήθειες. Θα πρέπει οι νομοθέτε να λάβουν μερίμνη για το ζήτημα αυτό. Οφείλουμε να το κάνουμε και θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένου στόχου χειροπιαστού, για να μα καθοδηγούν σε όλον τον χώρο των μεταφορών. Υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει σε όλε τι πόλει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Transport for London, ε, λογοχαρητερία αυτή που ασχολείται με τις συγκοινωνίε στο Λονδίνο, έχει ένα μεγάλο σχετικό πρόγραμμα. Το είπαν και άλλοι εδώ ε, για την εκπροσώπηση των γυναικών. Χρειάζεται να εκπροσωπούνται γυναίκε σε όλα τα επίπεδα. Και για πολύ καιρό, επειδή εργάζομαι εδώ και χρόνια στον τομέα των μεταφορών, στι θέσεις ε, management, τις ανώτερες, όσοι είναι senior manager, υψηλά στελέχη των επιχειρήσεων και των εταιριών σπανίω είναι γυναίκε. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με ε, εθελοντικά μέτρα. Πρέπει να υπάρξει κάποια υποχρεωτικότητα, κάποια δεσμευτικότητα. Χρειάζεται λοιπόν πραγματική δράση. Δράση από τους συμμετέχοντες στον τομέα των μεταφορών και όχι απλώς από το κέντρο προς τα έξω. Ευχαριστούμε, κύριε Άντροσαν. Κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η πρώτη ομιλήτρια από την Επιτροπή Γυναικών. Εγώ νόμιζα ότι είναι κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Γυναικών και Μεταφορών. Δεν το πήραμε είδηση μέχρι τώρα. Και θέλω να πω ένα θέμα αρχής και προς το πάνελ. Εμείς ε, γυναίκες έχουμε και μια ίδια αντίληψη για το πώς προωθούμαστε. Δηλαδή δεν θα μας προωθούν κάποιοι επειδή δεν έχουν άντρες. Ε, έχουμε λειψανδρία στις μεταφορές για φέρτε γυναίκες. Δηλαδή θέλετε να προσελκύσετε, να δελεάσετε, η γερμανική καμπίνα, ε, τις γυναίκες να πάνε στις μεταφορές. Ελπίζω να το καταλάβουν οι γυναίκες ότι ε, θέλουν να τους προσελκύσουν κάποιοι, να τους δελεάσουν σε ένα κλάδο που δεν μπορείς να βγάλεις το ψωμί σου που ε, δεν αποφέρει, δεν επικερδίζει και επειδή δεν πάνε άνδρε να φέρτε τι γυναίκε. Αυτό είναι πρόθεση των γυναικών. Αυτό δεν ε, εννοείται πρόθεση των γυναικών. Επειδή ε, έχουν, το έχουν βάλει στα πόδια ήδη άνδρες από εκεί. Ακούσαμε για του οδηγού φορτηγών και πώ έχει η κατάστασή του. Όποιο έχει την παραμικρή ευκαιρία να εργαστεί κάπου αλλού και να βγάλει λεφτά, δεν θα κάτσει να είναι οδηγό φορτηγού. Γιατί να πάει η γυναίκα και θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είμαι μόνη από την Επιτροπή Γυναικών, λέει η κυρία Νόχελ, και να το πω και στους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων. Εμείς δεν είμαστε εκεί μια μάζα που θα γεμίσει ε, ε το χώρο όταν λείπουν ε, οι άνδρες και όταν επιστρέψουν θα μας διώξετε. Βλέπετε τι γίνεται στον πόλεμο, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα και ακόμα και αεροπλάνα πετάνε. Ε, αλλά όταν δεν τις χρειάζονται ε, είναι άχρηστες. Χρειάζεται μια προσέγγιση αρχής και αυτό το βλέπουμε στην Επιτροπή Γυναικών. Το ξέρετε αυτό το αυγό, το σοκολατένιο που, το ανοίγεις και έχει μέσα ε, ένα παιχνίδι αν είναι κορίτσι και αγοράσει ένα τέτοιο αυγό, ε, δεν πρόκειται να βρει αυτοκινητάκι μέσα. Πάντα ε, είναι ε, μια κούκλα. Αν είναι κόκκινο ή ροζ το αυγό και αν είναι καφέ που είναι για γόρια, είναι αυτοκινητάκι. Και μετά ερχόμαστε και απορούμε. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα, θα μπορούσαν να είναι και στον κλάδο των μεταφορών, αλλά βλέπουμε συνέχεια ε, τις γυναίκες να υποβαθμίζονται, να υποβιβάζονται. Ε, και, και στην ε, Βαβαρία έχουμε μια πανηλήθεια παροιμία που λέει οι γυναίκες και τα κομμένα λουλούδια δεν έχουν καμία θέση σε ε, ένα πλοίο. Φανταστείτε, άκουσον, άκουσον, ωραία παροιμία. και Πραγματικά αυτό είναι αξιοπρεπέ για εμά τις γυναίκες που μας λέτε ότι έχουμε λιψανδρία φέρτε γυναίκες. Οι γυναίκες μπορούν ε, να κάνουν τα πάντα, μπορούν να προωθούνται παντού γιατί έχουν τα προσόντα και τις δεξιότητες και όχι επειδή ε, δεν έχουμε δυναμικό. Για τις γυναίκες είπατε ότι δεν μπορούν οι γυναίκες να οδηγούν τη νύχτα, την νυχτερινή εργασία. Οι νοσηλεύτριες κάθε νύχτα ξέρετε τι κάνουν στα νοσοκομεία. Και βεβαίω θα πρέπει αυτό να συνάδει με την οικογενειακή ζωή, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ δύσκολο τελευταίο. Αλλά ως Επιτροπή Γυναικών τόση ώρα μιλούν πρόσωποι της Επιτροπής Μεταφορών. Τελειώνοντας λοιπόν να πω ότι η προώθηση των γυναικών δεν σημαίνει κλείνω τρύπες σημαίνει έχουμε γυναίκες τις οποίες αντιλαμβανόμαστε ως ικανές ε, ε, και τις αναγνωρίζουμε για όλο τον κλάδο και τις τιμούμε. Και πρέπει να βελτιωθεί και η αμοιβή, γιατί οι γυναίκες έτσι και αλλιώς υπο, ε, αμείβονται. Ε, γυναίκες σε χαμηλόμιστες θέσεις έχουμε αρκετές, δεν χρειαζόμαστε άλλες. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Περιμένουμε όντως ε, και εμείς από την πλευρά μας συγκεκριμένε προτάσεις από την Επιτροπή των Γυναικών και ήταν καλοδεχόμενες για να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η Μαρία Νόχελ με κάλυψε πολύ. Εγώ δεν είμαι μέλος στην Επιτροπή Γυναικών αλλά υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα, όχι μόνο στις μεταφορές, αλλά πού χρησιμοποιούνται οι γυναίκες. Και ε, ακούστηκε ο κοινωνικός ρόλος των γυναικών, είναι μεγάλο πρόβλημα για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, όχι μόνο για τις μεταφορές. Η εικόνα της γυναίκας είναι αυτή, ότι να είναι σπίτι της, να κάνει παιδιά και τέτοια πράγματα. Ποια ισότητα. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες ε, είναι πιο πολύ στα κοινωνικά επαγγέλματα και οι άνδρες στα τεχνικά επαγγέλματα. Από το σχολείο αρχίζει αυτή η νοοτροπία. Χρειάζεται αλλαγή στα μυαλά. Ε, να ενισχύονται και οι γυναίκες και τα κορίτσια και τα γόρια σε όλους τους τομείς να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι τους ε, αρέσει, τι τους ταιριάζει και ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η φύλαξη των παιδιών. Πώς να πάει μια γυναίκα να δουλέψει όταν δεν ξέρει τι να κάνει τα παιδιά της, σε ποιο παιδικό σταθμό ε, είναι η σωστή φύλαξη των ε, παιδιών από επαγγελματίες με προσόντα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών δεν είναι ελκυστικό ο τομέα των μεταφορών, το ξέρουμε. Πρόσφατα μίλησα με κάποιον από μια μεταφορική εταιρεία. Ε, Νέου δεν βρίσκει ούτε άνδρε ούτε γυναίκε. Ούτε φιλικό προ την οικογένεια είναι το επάγγελμα. Ούτε η αμοιβή είναι ελκυστική. Γιατί να πάει ο άλλο να γίνει οδηγό σε φορτηγό, άνδρα ή γυναίκα. Γιατί να το κάνει αυτό στον εαυτό του, να δουλέψει σε αυτό το κλάδο. Αφήστε που και η ποιότητα τη δουλειά δεν είναι πάρα πολύ ελκυστική. Γιατί να αναζητήσει δουλειά, θα βρει αλλού ε, πολλά πρέπει να γίνουν, ε, ανεξαρτήτως αν είναι αυτό για τις γυναίκες ε, θέμα ή θέμα εργασιακό. Ο Στόχος θα πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξη. Βεβαίως οι γυναίκες είναι παντού σημαντικές, στα τεχνικά, στα κοινωνικά επαγγέλματα, αλλά και οι άνδρες. Γι' αυτό θα πρέπει συγκεκριμένα μέτρα να υιοθετήσουμε για όλους, άνδρες και γυναίκες. Και να είναι ελκυστικό το επάγγελμα και να αξίζει τον κόπο και να βγάζει και λεφτά όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στρέφομαι πλέον στις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στο πάνελ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές. Πώς να συνδυαστούν τον επαγγελματικό ιδιωτικό βίος, ποιότητα της εργασίας. Το είπατε και εσείς κύριε Μπαχ διάθεση να προσελκύσουμε τις γυναίκες σε ένα τομέα που αυτή τη στιγμή δεν είναι κερδοφόρος και πώς θα ξεκινήσει αυτό την πανεπιστημιακή παιδεία, τη σχολική εκπαίδευση. Έκκληση προς τις γυναίκες για να ε, εργαστούν σε αυτό το τομέα. Ποιότητα της εργασίας και πραγματικές απαντήσεις ε, χρειάζονται εδώ, αλλά γιατί τέθηκαν πραγματικές ερωτήσεις. Μας το είπε και ο κ. Βάντεν Κάμπ. Θα υπάρξουν αποσωστώσεις στην Ένωση. Διότι υπάρχει η ποσόστοση ισότητα στις διάφορες χώρες πλέον. Εάν υπάρξουν ποσοστώσεις, τι θα γίνει με τις εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν, ιδίως στον κλάδο των μεταφορών. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμη και στις ε, επιχειρήσεις σήμερα, το μερίδιο της μισθολογικής ισότητας η, η ίση εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τη εταιρεία μα οδηγεί πάλι να αναρωτηθούμε πού είναι οι γυναίκε σε θέσει ευθύνη. Προ τα κοιτίνουμε τελικά ή όχι. Όλα ουσιαστικά ακούστηκαν λίγο πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά μεταξύ μα στην παρουσίασή σα μιλήσατε για τι βίες συμπεριφορέ κατά των γυναικών. Και αυτό θα πρέπει να προσελκύσει την προσοχή τη Ευρώπη. Είναι πραγματικά θέμα επί της ουσίας αυτό. Οι μορφές βίας συμπεριφοράς κατά των γυναικών, παρενόχληση, ε, εκφοβισμός, σεξιστική παρενόχληση πολλές φορές η βία συμπεριφορά. Είδα μια μελέτη πρόσφατα που δείχνει ότι πολλές γυναίκες που εργάζονται στις συγκοινωνίες έχουν δεχτεί επίθεση τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους. Μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Και αν το συνδυάσουμε με τις βίες συμπεριφορέ, η βία κατά των γυναικών στις δημόσιες συγκοινωνίες είναι φρικτή. Φρικτή. Είπατε ότι οι γυναίκες παίρνουν περισσότερο τα μέσα συγκοινωνίας. Οκ, okay, ναι, συμφωνώ. Αλλά είδα μια μελέτη από ένα Ινστιτούτο που εδράζεται κυρίως στη Γαλλία, στο Παρίσι, και λέει 100% των γυναικών 100% των γυναικών που παίρνουν τι δημόσιες κοινωνίε, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους έχουν δεχθεί παρενόχληση στα μέσα δημόσιων μεταφορών από σεξιστική συμπεριφορά. Αυτό είναι πρόβλημα τη ουσία. Αυτά. Λοιπόν, να σας δώσω τον λόγο. Λυπούμε που δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα Μπορέσετε να μας στείλετε και γραπτές απαντήσεις μέσω mail αν θέλετε και αν δεν αρκούν τα δυόμιση λεπτά για τον καθένα και την καθεμιά σας. Να ξεκινήσουμε με εσά. Πάμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις στα γερμανικά γιατί μου ετέθησαν ερωτήματα από δύο γερμανόφωνες ε, βουλευτίνες. Φυσικά ε, δεν άκουσα ε, τη γερμανική μετάφραση για το αν μίλησα για δελεάζω ή προσελκύω. για τους νέους μίλησα και για τις γυναίκες. Και είπα ότι θα πρέπει να κάνουν πιο ενδιαφέροντα τον τομέα των μεταφορών και μιλούσα ιδιαίτερα για την εσωτερική ναυσιπλότητα, πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα του τομέα. Δεν ε, είπα ότι θα πρέπει να δελεάσουμε εμεί εξωτερικά, αλλά ίδιο ο τομέα πρέπει να, γίνει πιο ελκυστικό για να μπορεί και του ε, ε, ασκούμενους ε, και τους νέους να τους προσελκύσει. Εδώ πολλές φορές όταν μιλάμε για μεταφορές περιοριζόμαστε, σκεφτόμαστε μόνο δικές μεταφορές. Εδώ ε, μιλώ όμως για την εσωτερική ναυσιπλοεία που ε, μπορεί να προσφέρει θέσεις εργασίας δεν μιλάμε μόνο για αυτούς που ζουν πάνω ε, στη φορτηγίδα, πάνω στο πλοίο, που άντρας, γυναίκα, που είναι ιδιοκτήτες του πλοίου, έχουν την ίδια κατάρτιση και κάνουν τις ίδιες δουλειές. Όμως η εσωτερική Πλοιά προσφέρει και θέσει εργασία σε υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει και πολλές δυνατότητες επιμόρφωσης, ε, περαιτέρω εκπαίδευσης. Επειδή υπήρξε αυτή πρόταση, ε, το αναφέρω, η πρόταση της Κομισιόν για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων πρέπει να γίνει στην Ευρώπη συνολικά. Επίσης, ε, αποκοινούμε τους κοινωνικούς εταίρους, προσπαθούμε τις σχέσεις εργασιακές, το ωράριο εργασίας, ε, να αναδιαμορφώσουμε τις σχετικές διατάξεις στην εσωτερική ναυσιπλοεία και θέλουμε να είναι όλο και πιο ελκυστικέ θέσει εργασία πάνω ε, στι φορτίες πάνω στον τομέα τη αστερικής ναυσιπλοεία και για τις γυναίκες, ε, ε, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε και στις γυναίκες εξειδικευμένε θέσει εργασία. Είναι ένας τομέας που πιστεύω ότι εδώ έχει μεγάλη σημασία η επιμόρφωση, η περαιτέρω κατάρτιση και, και εκεί σκοπεύουμε. Έγιναν και κάποιες, κάποια άλλα σχόλια. Είπατε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία ε, για το, με το πρόγραμμα σπουδών. Μας ενδιαφέρει και μας στην τομέα της εκπαίδευσης ε, να αναφέρουμε, ε, να προωθήσουμε αυτά τα επαγγέλματα και σε ό,τι αφορά τη νέα πρόταση Κομισιόν για την, τα επαγγελματικά προσόντα. να μπορεί κάποιο που έχει χρηματίσει στο πλοίο πάνω και έχει κάνει κάτι να μπορεί μετά να βρει μια θέση στη στεριά. Γενικά υπάρχουν πολλές προτάσεις, πολλές ενδιαφέρουσες λύσεις και προσεγγίσεις. Και σίγουρα υπάρχουν πολλέ γυναίκε που ενδιαφέρονται για τα τεχνικά επαγγέλματα, ε, στην εφοδιαστική για παράδειγμα, και μπορούν να απασχοληθούν ε, στο μέλλον. Βέβαια, στην εσωτερική ναυσπλά σίγουρα υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και αυτό το πρόβλημα προσπαθούμε μαζί με του κοινωνικού εταίρου να το λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τίλινγκ έχει τώρα το λόγο. Να ξεκινήσω απαντώντας στην ερώτηση του κυρίου Βάντεν Κάμπ. Πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να υπάρξει ισότητα στις μεταφορές. Δεν είναι το πρόβλημα να έχουμε 50% αντρες γυναίκε στον κλάδο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί ο καθένας να κάνει την επιλογή αν θέλει με τρόπο ισότιμο. Στον κλάδο των μεταφορών αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιλογές προσφέρονται στους άντρες και όχι στις γυναίκες. Αυτός είναι ο λόγος. θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλε προποθέσει ώστε να υπάρχει ίση δυνατότητα επιλογής και ίση συμμετοχή. Λύσεις. Βεβαίω, στην ETF πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες, διότι η... τα ήπια μέτρα βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο στην Ευρώπη. Η επιβολή του νόμου, ειδικά του τομέα μεταφορών στον οποίο εργαζόμαστε, ξέρουμε τι σημαίνει. Είναι αδύναμη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι λύσεις μπορεί να υπάρξουν. Νομικό πλαίσιο για να δούμε τελικά, και με συγχωρείτε που θα το πω, το ζουμί είναι οι εταιρείε και οι χώροι εργασία. Εκεί πρέπει να δούμε την επιβολή του νόμου. Εκεί να δούμε αν οι εταιρείε καταρτίζουν προγράμματα ισότητας τα οποία να αφορούν την εκπροσώπηση στα υψηλότερα ε κλίμακα της εταιρεία και το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται και να είναι, ένα εργαλείο, να που λειτουργεί. Και επίσης πολλές εταιρείε δεν ε, οργανώνουν αρκετό διάλογο. Το έθεσαν και άλλοι ομιλητές. Ο κοινωνικός διάλογος και πάλι εννοώ ότι σε κάποια κάτι μέλη της Ευρώπης δεν υπάρχει περίπτωση να συσταθεί η συνδικαλιστική οργάνωση εντό μια εταιρεία. Το να μιλήσει για ισότητα φύλου κανεί είναι ακριβώ θέμα κοινωνικού διαλόγου. Έτσι πρέπει να δούμε λόγου χάρη πώ ήταν οι βάρδιε ανδρών και γυναικών περίπου ισότιμε. Εάν δεν υπάρχει κάποιο επικεφαλή στην εταιρεία που να ασχολείται με τα θέματα αυτά, πού να πάει να το συζητήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι πραγματικά συμφωνώ απολύτω, οι γυναίκε δεν πρέπει να γίνουν οικονομικό θύμα αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστούμε κυρία Τίλινγκ. Κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ. Πολύ πλούσια συζήτηση. Πραγματικά χρειαζόμαστε σφαιρική προσέγγιση δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Είναι σαν να προσπαθήσει κανεί θα πρέπει κανείς να δει το παλιό τρόπο που χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούσε και ο πατέρας μου για τις ε, που έπρεπε να τις πατήσεις ξανά και ξανά για να βγουν στο χαρτί. Την πρώτη δεν έπιανε, τη δεύτερη κάτι γινόταν, την τρίτη έβγαινε. Ε, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να αναζητούμε μαγική λύση. Χρειάζεται κοινωνικός διάλογος, χρειάζεται κοινωνικός διάλογος μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων, των κοινωνικών φορέων, δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε ένα μόνο επίπεδο, ευρωπαϊκό ή εθνικό ή επιχειρήσεων κ.ο.κ. Πρέπει όλα τα επίπεδα να βρισκούνται σε συνεργασία μαζί μεταξύ του. Και αυτά που είπε η κυρία Γιάλα Σέντερ, αν και έφυγε από την αίθουσα δυστυχώ, θα τη απευθυνθώ διμερώ για να τη πω για τα στατιστικά στοιχεία. Μπορεί να ακούγονται κάπω στεγνά και βαρετά τα στατιστικά στοιχεία, όμω οι αριθμοί και τα στοιχεία χρειάζεται να μελετώνται όπω από την αρχή. Θα φροντίσω να τη πω γιατί. Ακόμη και για τι μεταφορές και τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Το θέμα είναι πώς τα βλέπουμε τα θέματα αυτά. Τι επιλογές κάνουμε, τι προποθέσει προσφέρουμε. Χρειάζεται η ισορροπία επαγγελματικού ιδιωτικού βίου, όπως είπατε κύριε Μπάκ. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, όχι μόνο για το σκοπιά του θέματος στενά, αλλά και για τα υπόλοιπα γενικότερα. Γι' αυτό στρέφομαι στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πολιτική ηθήνοντες. Πιστεύω ότι μπορείτε να κάνετε πολλά, αλλά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Θα ολοκληρώσω ένα άνδρα τη σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω καταρχά να απαντήσω στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Μπαχ για το πιλωτικό πρόγραμμα για την ληστικότητα των μεταφορών. Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω ε, κάπως γιατί προς το παρόν δεν έχουμε πολύ οριστικά αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σύντομης διάρκειας, ε, μόνο κάποιους μήνες διαρκεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα από ε, μια εταιρεία συμβουλών πάρα πολύ ε, καλή που πρώτα έκανε απογραφή των υφιστάμενων εργαλείων και έπειτα πέρασε στη φάση συλλογής στοιχείων από έρευνες σε νέους άνδρες και γυναίκες, τους οποίους ε, ρώτησε διάφορα πράγματα για να δει πώς αντιλαμβάνονται και τι προσδοκούν από τον τομέα των μεταφορών. Είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση, δεν έχουμε τα αποτελέσματα. Από ό,τι φαίνεται πάντως δεν είναι και τόσο κακή η αντίληψη που έχει ο κόσμος ε, και αυτή που περιμέναμε να έχει ε, για τις μεταφορές, αλλά τα αποτελέσματα τα έχουμε πολύ γρήγορα, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Η κυρία Γιάλα Σέντελ δεν είναι εδώ, οπότε επειδή εξέφρασε τη λήψη που δεν ήταν παρούσα Επίτροπος, δεν σημαίνει ότι δεν την ενδιαφέρει το θέμα. Το αντίθετο έχει δείξει μέχρι τώρα στάση και πρωτοβουλίε που έχει αναλάβει σε ό,τι αφορά το ότι υπάρχουν λίγες θέσεις και πάρα πολλές γυναίκες με πτυχίο και άρα πώς να καλύψουμε και θέσεις που, ε, με γυναίκες που δεν έχουν πτυχίο θαύματα δεν μπορούμε να περιμένουμε στον τομέα αυτό. 3% ε, έχουμε μόνο μηχανοδηγούς γυναίκες. Δεν θα φτάσουμε στο 50% ποτέ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, εκεί μπορεί να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Για τα ασφαλή πάρκη, τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης, ε, Υπάρχει μια πιο ευρία διάσταση. Στις ε, επαφές που είχαμε, το πρόβλημα είναι περισσότερο οι υγειονομικές εγκαταστάσεις ε, και αυτό αφορά γενικώ τους ε, χώρους εργασίας. Σίγουρα είναι όμως ένας ακόμα παράγωνα που αποτρέπει τις γυναίκες, παραδείγματος χάρη ασφαλή χώρου χώρους στάθμευσης, στις οδικές μεταφορές. Θα δούμε σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε, την πλατφόρμα για την αλλαγή, τι πρακτικές θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και τι χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, ίσως μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων. αυτά είναι υποδιερεύνηση. Πολύ γρήγορα τώρα για τις ποσοστώσεις. Άκουσα αυτό που με ρωτήσατε. Το σκεφτόμαστε. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι είναι άκρος πολύπλοκο το ζήτημα. Γιατί σε κάθε τρόπο μεταφράζει διαφέρει η κατάσταση. Και βέβαια, στον προβληματισμό μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλα ζητήματα, Όπω είναι οι οι στόχοι. Οι δείκτε επίσης είναι ένα θέμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να σκεφτόμαστε πάνω στο θέμα. Είναι δυναμική ολη η διαδικασία. Στην αρχή είμαστε ακόμα λίγη υπομονή λοιπόν και λίγη κατανόηση γιατί Μόλις ένα χρόνο ε, έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, για να ολοκληρώσουμε, ε, θα δώσω το λόγο για ένα λεπτό στον εισηγητή μας, βέβαια, τον κύριο Νίλσεν. Ναι, πράγματι ένα λεπτό ε, θα χρειαστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ακούσαμε διάφορες απόψεις με τις οποίες συμφωνούμε και υπάρχουν και κάποια συμπεράσματα. Ότι δηλαδή ο κλάδο πρέπει να είναι ελκυστικό, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και τα κοινωνικά ζητήματα. Πώ ε, γίνεται δουλειά, τι προσφέρουν οι εταιρείε. Επομένω πιστεύω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το συνδέσουμε με άλλα ζητήματα που μας απασχολούν στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή Απασχόλησης βέβαια, διότι η χώροι εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλη για όλου. Αν εκεί δεν ε, καταφέρουμε ε, κάτι καλύτερο, θα χάσουμε την ευκαιρία να έχουμε έναν ε, καλύτερο τομέα που θα είναι ελκυστικός και για άντρες και για γυναίκες. βλέπω και σε νέες ακροάσεις, ίσως να δούμε κάποια καλά παραδείγματα και να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα παρανόητα να τα διαδώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε και τον κύριο Νίλσεν. Φυσικά θα συνεχίσουμε έργο αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή Γυναικών και την Επιτροπή Απασχόληση. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, όλες και όλους, που μας κατήφθηναν σε συγκεκριμένε πίστες για να βρουν οι γυναίκες αύριο τη θέση τους στην αγορά εργασίας των μεταφορών. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε 3 η ώρα το μεσημέρι για να συνεχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής Μεταφορών. Καλή όρεξη και ευχαριστή πρόεδρος τους διερμηνείς. Που φαντάζεται ότι είμαστε κι εμείς πολύ ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τα θέματα των γυναικών στις μεταφορές.